Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθίστε, παρακαλώ, ήσυχα και χωρίς συνομιλίες. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε την ημερησία μας διάταξη. Σήμερα το πρωί έχουμε στη θέση μας και το απόγευμα συνεδρία της Επιτροπής. Φανή, Έχουμε λοιπόν συνεδρίαση της Επιτροπής πρωί και απόγευμα, υπεπισμένη ότι θα έρθουμε και πιο αθρώοι στα έδρανα σιγά σιγά, ως συνήθως. Ως συνήθως δε έχουμε και διαδικτυακή μετάδοση της συνεδριάσεως. Και Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση στο πρόγραμμά μας για να μην έχουμε προβλήματα. Τα δύο κομμάτια της συνεδρίας θα έχουμε χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο τμήμα θα ασχοληθεί με μια γενική συζήτηση της προτάσεως εκθέσεως του Σαλβαδόρ και στο δεύτερο, α, το πρώτο, το πρώτο θα μας πάει μέχρι τις 10 και 4. Το πρώτο τμήμα. Μετά θα αρχίσει η δεύτερη φάση της συζήτησης όπου θα έχουμε όχι οριζόντια, αλλά εν πάση περιπτώσει μια συνολική θα έλεγα θεώρηση της κατάστασης, οριζόντια κάπως κατανομή δηλαδή, αν όχι μέκή όχι το τομέακη και λιγότερο χρόνο για συζήτηση και έτσι το απόγευμα με το τρίτο τμήμα μπορούμε να συζητήσουμε διάρκειες, δομές και ούτω καθεξής μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από τις 5 και μετά και κλεισμένο των θυρών θα γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών που θα προετοιμάσει την προσεχή συνεδρίασή μας. Ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Ε, γρήγορη και αποτελεσματική, όπως πάντα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Και γι' αυτό προχωρώ αμέσως τώρα στο πρώτο τμήμα της συνεδριάσεως που θα κάνει όπως πάντα, που θα εισαγάγει όπως πάντα ο Σαλβαδόρ. Γενική λοιπόν ώρα της έκθεσής του. Και στη συνέχεια με τη σειρά οι ομάδες εκπροσωπούμενες από τους συντονιστές τους θα κάνουν τα σχόλιά τους για το Γενικό Τμήμα με την συνηθισμένη σειρά πλήν της εξής εξαιρέσεως ότι μου ζητήθηκε το ΕΛΚ να μιλήσει τελευταίο, δηλαδή ο συντονιστής του ΕΛΚ να είναι ο τελευταίος ο οποίος θα λάβει το λόγο σε αυτή τη σειρά, ο κ. Ράμαρ Μπέγκερ, ακριβώς επειδή έχει τον εισηγητή το ΕΛΚ, βέβαια ο εισηγητής είναι εισηγητής όλων μας ε, φασών και παντών, αλλά εν πάση περιπτώσει ας είναι τελευταίος ο εισηγητής του ΕΛΚ που θα λάβει το λόγο στη σειρά. Δεν θα ήταν πολύ καλό να μιλήσει πρώτα ένας εισηγητής από το ΕΛΚ και μετά ένας συντονιστής από την ίδια ομάδα. Γι' αυτό κάναμε αυτή την αλλαγή στη σειρά. Παρακαλώ λοιπόν τώρα τον Σαλβαδόρο, ο οποίος έχει θέση του 10 λεπτά, εάν τα χρειάζεται. Αν δεν τα χρειάζεται δεν πειράζει, τόσο καλύτερο. Και έτσι κερδίζουμε χρόνο όλοι. Και αφού ακούσουμε βέβαια τους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες, ανοίγει η συζήτηση για όλους. Έχουμε χρόνο για τη γενική συζήτηση μέχρι τις 10 και 4. Παρακαλώ, Σαλβαδόρ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και 6 μήνες ε, χρησιμοποιώ πέντε λεπτά στι παρουσιάσει μου, επομένω ε, θα συνεχίσω μετά τα συνηθισμένα μου λεπτά, δεν χρειάζομαι τα παραπάνω. Θα αναφέρω εδώ διάφορους, ε, η κυρία Πολύνια Στράση, ο Χούλη Ροντρίγκε, η η και η Λουσία Γρογιοκάνου. Και κατόπιν Φάνη, Νικόλ και Ανά Μαρία από το ΕΛΚ ε, που εργάστηκαν ε, όλους αυτές τις μήνες πολύ σκληρά για να μπορέσω να σας παρουσιάσω μια έκθεση. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την επαγγελματικότητά τους για την αφοσίωσή τους ε, και φυσικά ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις συζητήσει όλους αυτούς τους μήνες, ε, συζητήσει των οποίων το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται σήμερα στο έγγραφο. Πρόκειται για ένα έγγραφο που καταρχήν προσπαθεί να αντικατοπτήσει μια συνένεση μεταξύ όλων των μελών αυτής της ειδική Επιτροπής και το δεύτερο είναι να πετύχουμε στην Ολομέλεια ψηφοφορία άνω των 500 ψήφων για να μπορέσουμε να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο για την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Η έκθεση αυτή, θα θυμάστε, αποτελεί μία σύνοψη, μια συνέπεια των εναποκείμενων συζητήσεων όλων αυτών των μηνών για τα διάφορα θέματα που συνιστούν τις δημοσιονομικές προοπτικές. Θέλω να σας πω ότι εμείς αναλύσαμε τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν εμβαθύναμε στην πολυπλικότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών των πολιτικών όπου χρειάζεται, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κάνουν οι αρμοδίες επιτροπές αυτού του Κοινοβουλίου. Εμείς ε, απλώς αναφέρουμε κάποιες πολιτικές ε, ενδείξεις ε, και μιλάμε για την δημοσιονομική διάσταση που είναι απαραίτητη για την πρόθεσή τους. Η μέθοδο εργασίας, μέθοδος εργασίας εκπονήσαμε τρία έγγραφα εργασία όλο αυτό το καιρό. Ένα για την Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία, ένα για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και κατόπιν για τα τεχνικά μέτρα που αφορούν τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, δομή, διάρκεια και ευελιξία. Αυτά τα έγγραφα εργασία μαζί με τη σύνοψη που εκπονήσαμε όταν ολοκληρώσαμε τις ε, συνεδριάσεις εργασίας αποτελούν τη βάση της έκθεσης. Βεβαίως, χρησιμεύσαν ε, και τα γραπτά σχόλια που έστειλαν οι διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά και τα μεμονωμένα σχόλια, καθώς και το feedback που είχαμε με τα εθνικά κοινοβούλια σε όλες τις περιπτώσεις. Ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο, αλλά δώσαμε, έχουμε αφήσει και πολύ μεγάλο χώρο σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, ακριβώς για να συμπεριλάβουμε κάθε πρόταση και αντίθετη θέση και τροπολογία που μπορεί να προκύψει από τις πολιτικές ομάδες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τροπολογιών θα έχουμε ως προθεσμία την 8 Ιουνίου και θέλουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση επί της οποίας θα συμφωνούν οι περισσότεροι. Καταρχήν, ε, για τη δομή έχουμε μία ανάλυση για τις ε, κύριες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον προϋπολογισμό για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Δεύτερον, αναλύονται αυτές οι προκλήσεις ανάλογα με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Προσθέμενης Αξίας, της αποτελεσματικής δαπάνης και του πιθανού αποτελέσματος που μπορεί να έχει ένας κοινοτικό προϋπολογισμός όταν ε, χρησιμοποιούνται άλλα είδη δημόσιων ε, κονδυλίων και καινοτόμα εργαλεία. Και νομίζω ότι έχουμε και το πιο πολιτικό τμήμα της έκθεσης που αφορούν τις προτεραιότητες της Ένωσης. Εγώ τις ε, ανέλησα ανέλησε τις κύριες ε, βασικές ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουμε την αηφόρο ανάπτυξη, την ευφυή ανάπτυξη. Έχουμε την πολιτική συνοχής, της πολιτικής μετανάστευσης ασφάλειας και ηθαγένειας και την εξωτερική πολιτική και θα προσθεθεί και μία παράγραφος που θα συζητήσουμε το απόγευμα για την χρηματοοικονομική διακυβέρνηση. Σε όλα αυτά πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο η στρατηγική για το 2020. Κάνω ορισμένε συστάσεις για την νέα για τη διάρκεια και για τους κανόνες ευελιξίας που θα έπρεπε να διέπουν τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και κάνουμε και μία δήλωση για τους απαραίτητους πόρους, το μέγεθος του προϋπολογισμού και ω ποιο βαθμό, ως ποιο σημείο οι νέοι διπόροι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή τη δήλωση. Ω οριζόντια θέματα τώρα, φυσικά αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και κυρίως στη στρατηγική την Ευρώπη το 2020 που θα πρέπει να είναι η κύρια πολιτική αναφορά των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά όχι Όλες ε, οι ε, ιστορικές πολιτικές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ε, αυτή τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και νομίζω ότι η δομή που προτείνουμε καθιστά ε, ιδιαίτερα ορατή αυτή τη στρατηγική. Προβάλλει αυτή τη στρατηγική όμως χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες διευκρινήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά στο πώς οι θεματικές ε, πρωτοβουλίες, τα flagship initiatives, ε, θα ποσοτικοποιηθούν από τη σκοπιά του προϋπολογισμού. Ακόμη δεν υπάρχει τέτοια ποσοτικοποίηση, πάντως η στρατηγική για το 2020 θα πετύχει αν είναι επαρκώς αξιόπιστη και αν χρηματοδοτηθεί σωστά μέγεθος του προπολογισμού. Είναι προφανές και αναλύεται στην ε, έκθεση ότι πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους από το 2014 και μετά. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί για τον προπολογισμό της Ένωσης και όλα τα σύμβανα του Συμβουλίου μας δείχνουν ότι το ίδιο θα ισχύει και τα επόμενα έτη. Αν ε, ε δεν υπάρξουν ε, νέοι πόροι για την χρηματοδότηση των πολιτικών της Ένωσης έχουμε αυτή την δυνατότητα με την χρήση των ίδιων πόρων. Ε, έχουμε το 1,23% του καθάριστου ε, κοινοτικού ε, χώρου προϊόντος. Ψηφίστηκε αυτό από το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και φυσικά γνωρίζουμε ότι τις δαπάνες θα πρέπει να τις αναδιαρθρώσουμε σε πάρα πολλούς τομείς και να, καταστήσουμε πιο να τις καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παγώσουν ε, οι κοινοτικέ δαπάνες, ε, αν τουλάχιστον θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά και των ε, πολιτικών μετά τη Λισαβόνα και αναφέρομαι κυρίως στις ανάγκες της πολιτικής συνοχής και της κοινή αγροτική πολιτικής. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι οι πολιτικές και χρηματοοικονομικές προκλήσεις τίθενται επιτάπητος. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί με σαφήνεια μέσω της κοινοτικής μεθόδους αντί της διακυβερνητικής προσέγγισης. Κατά την άποψή μου ε, αυτή την ε, κλίση παίρνουν τώρα τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ίσως επειδή έχουμε και τον επίγοντα χαρακτήρα της οικονομικής κρίσης, όμως εγώ νομίζω ότι αυτή τη μέθοδο πρέπει να ακολουθήσουμε και υπάρχουν σαφή πολιτικά μηνύματα σε αυτήν την έκθεση για να επιλέξουμε την κοινωτική μέθοδο έναντι της διακυβερνητικής προσέγγισης. Αυτά εισαγωγικά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μας περάσει όπως είπαμε το ΕΛΚ τελευταίο, και ως εκ τούτου και αναπάντεχα πρώτα, πρώτοι οι σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Σαλβαδόρ. Το έχω πει και πριν, αλλά ιδιαίτερα πιστεύω ότι πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να συνηθίσουμε τη δουλειά μας. Ε, η έκθεση του Σαλβαδόρ, τον ευχαριστώ πολύ, έχει ακούσει με προσοχή τα όσα είχαν να πούνε και τα μέλη της Επιτροπής και οι διάφορες ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αποτελεί, αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την περαιτέρω δουλειά μας η έκθεση του Σαλβαδόρ. Πλην όμως, γιατί ξέρετε, συνήθως υπάρχει και το αλλά. Πλην όμως, ο κίνδυνος, εν προκειμένου, με τη στάση και τις προσπάθειες του Σαλβαδόρ είναι ότι μπορεί να χαθούμε σε μια ε, προσπάθεια να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαθιστή, δηλαδή να γίνουμε πιο συντηρητικοί με την έννοια ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προασπίζουμε τα όσα έχουμε ήδη ως κεκτημένα, αλλά δεν έχουμε μεγαλύτερο όραμα για το μέλλον. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε πάνω από όλα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε όλοι, ζήσαμε όλοι μαζί το, τη μάχη για τον προϋπολογισμό, τις, ε, τη στάση και τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν, τις συζητήσει όχι μόνο για τον προϋπολογισμό του, του 2011 αλλά και για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές επεδοκρατών μελών, για ε, παγώματα, περικοπές, ακόμη και δραστικές περικοπές που μας περιμένουν. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Πρέπει να επιδείξουμε σαφή πολιτική βούληση για μια πιο φιλόδοξη πολιτική ατζέντα για ένα πρόγραμμα πολιτικό πιο φιλόδοξο και αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε πάνω από όλα. Και ως εκ τούτου, σε, ως προς αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε την έκθεση του Σαλβαδόρ πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει οικονομική κρίση. Τι συνέβησε για τον προπολογισμό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δεχθούμε το επιχείρημα τη λιτότητα άνευ ε, εταίρου. Δεν πρέπει να πούμε ότι είναι αναπόδραστο το αποτέλεσμα τη λιτότητα λόγω τη οικονομική κρίση. Πρέπει να βρούμε επιχειρήματα για να το ε, αντικρούσουμε φυσικά το επιχείρημα αυτό και από τι συζητήσει και τι προηγούμενη εβδομάδε, θα ήθελα να επισημάνω ότι ίσω θα μπορούσαμε επί τη ευκαιρία ή μέσα συνθήκε αυτέ, να προβούμε σε μια ανάλυση των εναλλακτικών. Τι συνέπειε θα είχε μια δραστική περικοπή στον προπολογισμό. Να αναλύσουμε τι συνέπειε, αυτές. Όχι μέσα στην έκθεση, αλλά χωριστά και σαν βάση για τι επιχειρηματολογίε που θα έχουμε να αναπτύξουμε. Και επίση θα πρέπει να αναλύσουμε τι συνέπειε επί των εθνικών προπολογισμών ε, τον αντίκτυπο, αν θέλετε, των εθνικών προπολογισμών μια πιο φιλόδοξη πολιτική. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη για να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα. Πρώτο σχόλιο λοιπόν, πρέπει να είναι πιο σαφή πολιτικά η κατάσταση για μα, να έχουμε πιο πολλά πολιτικά οράματα, φιλοδοξίε, να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα για το μέλλον της Ευρώπης και πάνω απ' όλα να αναζητήσουμε και να βρούμε τα επιχειρήματα αυτά τα οποία θα στηρίξουν αυτό το μέλλον της Ευρώπης. Και δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σαφές πάντοτε το τι προσθέμενη αξία έχει να προσφέρει η Ευρώπη ε, με βάση κάποιες προτεραιότητες. Αυτό πρέπει επίσης να πράξουμε. Είναι άκρο σημαντικό για μας και εδώ συνδέω και με την ε, έκθεση Παλτσάνη και τον προπολογισμό για το 2012 ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, θέσει εργασία, στην ανάπτυξη και τι επενδύσει, και αυτά είναι τα επιχειρήματα, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό για επενδύσει κλειδιά που θα καταστήσουν απόλυτα λειτουργική την εσωτερική αγορά, που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να είναι πιο ενωμένη και στι μεταφορέ, χάρη σε επενδύσει και στι μεταφορέ και στην ενέργεια και σε όλα τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πραγματικά την ευκαιρία που μας προσφέρει αυτό το πλούτο των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Όχι μόνο 27 κράτη-μέλη, πρέπει να κοιτάμε αυτό, αλλά 500 εκατομμύρια πολίτες. Και πρέπει επίσης να ε, συμπληρώσουμε και μια πολύ σημαντική προοπτική που δεν βλέπω ξεκάθαρα στην ε, έκθεση του Σαλβατόρ την αηφορία ή βιωσιμότητα, κάτι το οποίο ε, συζητούμε μακρόν για λόγους περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς. Αυτό είναι ένας ε, παράγοντας, μία έννοια την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ε, και αν δεν μπει στην έκθεση δεν θα είναι ίσως δυνατόν να προστατεύσουμε τις προτεραιότητές μας ως προς τις πράσινες επενδύσεις ή την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν αυτές, αλλά η αρχή της αηφορίας δεν εμφανίζεται αρκετά ξεκάθαρα μέσα στην έκθεση. Τρία πράγματα λοιπόν για να συνοψίσω. Πρέπει να πράξουμε. Πρώτον, πρέπει να διατυπώσουμε πολιτικά το πολιτικό όραμα της Ευρώπης, για το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να μιλήσουμε και να βρούμε λύσεις για επενδύσεις και πρέπει να συμπληρώσουμε την έκθεση με την αρχή της αηφορία. Τέλεια, λέει η πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε λεπτά. Κάρλ, τώρα. Ευχαριστώ. Καταρχά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σαλβαδόρ για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία ασφαλώς και αποτελεί ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης των συζητήσεων. Είναι πραγματικά μεγάλη η πρόκληση που αντιμετωπίζετε. Έχετε φιλοδοξία να συγκεντρώσετε 500 ψήφους ε, στην Ολομέλεια. Σωστή μεν, ωστόσο, για να το πετύχετε αυτό, φυσικά μπορεί να καταλήξετε με αυτό που μόλις μας είπε ο Γιώραν, ε, τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτό σημαίνει η Ευρώπη. Μιλάμε πολύ για αλλαγή και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, αποστέλει τέτοια μηνύματα εδώ και καιρό ότι πολλές είναι οι μελλοντικές προκλήσεις, καταρχάς οι οικονομικές, αλλά και το γεγονός ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το περιβάλλον χρειάζεται πιο πολλές επενδύσεις, ότι έχουμε αυτή τη στρατηγική το 2020 που είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν έχει ακόμα την κατάλληλη χρηματοδότηση για να στεχθεί με την επιτυχία που χρειάζεται και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, πολλές προκλήσεις ακόμα. Είναι λίγο κοινικό το γεγονός, φαντάζομαι, ότι η απάντηση στην έκθεση του Σαλβαδόρ είναι πιο πολλά χρήματα. Ε, ναι μεν, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά χωρίς πολλά χρήματα, πιο πολλά χρήματα, αλλά το θέμα είναι από πού θα πάρουμε τα χρήματα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αν θα συνεχίσουμε με, βάση την έκθεση αυτή, ε, θα, αυτό θα σημαίνει ότι θα αυξάνονταν πάρα πολύ ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε. Αυτό φυσικά είναι και θέμα αρχή. Κάποιοι μπορεί να είναι υπέρ, κάποιοι είναι και κατά. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλουμε. Το θέμα είναι και το τι είναι εφικτό. Και στο σημείο αυτό δεν είμαι βέβαιο κατά πόσο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουμε και καλωσορίζουμε την έκκληση για πιο πολλά χρήματα για την έρευνα, την ανάπτυξη, την τεχνολογία, για τους στόχους που έχουν τεθεί στην στρατηγική της 2020, αλλά εξακολουθώ να ρωτώ πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση. Αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν υπάρχουν αρνητικές προτεραιότητες στην έκθεση αυτή. Και τι εννοώ λέγοντας αρνητικές προτεραιότητες, οικονομίες. Ξέρω ότι το θέμα της οικονομίας και της εξοικονόμησης ε, πόρων ε, το αποφεύγουν γενικά οι πολιτικοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα αναγκαστούμε να ορίσουμε κάποιες αρνητικές προτεραιότητες και νομίζω ότι καλό θα ήταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει κάποιες αρνητικές ε, προτεραιότητες για να γίνει ακριβώς η επανακατανομή των κονδυλίων για να χρηματοδοτηθούν τα χρήματα τα οποία ζητάει ο Σαλβαδόρ. Γιατί Φυσικά τα πήγε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το πού θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χτες και ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Κοινοβουλίου είπε ότι αν είναι να αρχίσουμε να κοιτάμε τις επικεφαλίδες θα πρέπει να υπάρχει ίσως μόνο μία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν θέλουμε πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό Ξέρω ότι ακούγεται κάπω ριζοσπαστικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού προσπαθούμε να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά το θέμα, α το εξετάσουμε και αυτό σαν ενδεχόμενο. Μα χαροποιεί το γεγονό ότι στην έκθεση αναφέρονται και οι ίδιοι πόροι, γιατί η ομάδα μα θέλει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, αλλά η όλη συζήτηση για τους ίδιους πόρους θα πρέπει να αφορά και νέους τρόπους χρηματοδότησης ε, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, όχι μόνο το να λέμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και να φροντίσουμε να μην καθυστερήσει δυστυχώ η συζήτηση στο Συμβούλιο, το οποίο δυστυχώ ήταν εύκολο. Καλωσορίζουμε το γεγονό ότι αναφέρεται και το θέμα των ε, ομολόγων και είμαστε κάπω διστακτικοί σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του ετέ. Εμεί θα προτιμούσαμε ένα πενταετέ μοντέλο και μια μεταβατική περίοδο Άρα στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Τέλος, συζητήσαμε πολλά θέματα επιπρόσθετης αξίας. Πολύ ωραία αυτή η έννοια της ε, προστιθέμενης αξίας και ταιριάζει σε τέτοιες εκθέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο ειλικρινείς μεταξύ μας όταν συζητάμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, γιατί κάποια πράγματα που αναφέρονται ω ε, στοιχεία που θα συνδράμουν στην προστιθέμενη αξία μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα από ό,τι ω σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Λεκύη Πρόεδρο. Οι δικέ μου ε, αντιδράσει ε, προ το παρόν είναι ότι οι αντιδράσει πάντα είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το ποιο είναι ο εισηγητής. Κάποιο βγαίνει και λέει ναι, να ορίσουμε αρνητικέ προτεραιότητε. Ναι, μα να βγει κάποιο πρώτο να μα πει ποιε είναι αυτέ οι αρνητικέ προτεραιότητε. Καρλ. Δεν το λέω αυτό μόνο στι άλλε ομάδες, το έχω πει και στη δική μου ομάδα, γιατί και, και εκεί φυσικά έχει τεθεί αυτή η απέτηση, η αξίωση. Ναι, μα πείτε μου εσεί ποια είναι η αρνητική προτεραιότητα, να τη συζητήσουμε, να την εφαρμόσουμε. Αλλά τώρα μόνο απλά να το αναφέρουμε δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε έτσι. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε η Χέλγα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση του Επιτροπού Έτλικερ αυτή την εβδομάδα ότι πρόκειται να κάνει τουλάχιστον μία συζήτηση για το, πυρηνικό, για το πυρηνικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον για το μέλλον χωρίς πυρηνικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, εγώ ως Ευρωβουλευτής είμαι υπέρ τέτοιων αλλαγών προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι λοιπόν ξεκινώ με μία ε, γενική πολιτική συνήθεια της Κυριακές, ε, ο Μπαρόσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαϊκοί ηγέτες ε, μιλούν για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, να λύσουμε όλα τα ενεργειακά προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να έχουμε ευφύ και συμπεριληπτική ανάπτυξη και τελικά όταν επανερχόμαστε στον προϋπολογισμό μας και στην καθημερινή μας συμπεριφορά, ε, είναι πάρα πολύ συντηρητικοί, δηλαδή θέλουν να κρατήσουν τα πράγματα πάνω κάτω ως έχουν. Και νομίζω ότι δεν είναι η πιο ευφύης πολιτική συμπεριφορά αυτή. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω από τη δική μας σκοπιά, τις δυνατότητες αποταμίευσης, εξοικονόμησης. Ε, για, σε σχέση με όσα γίνονται στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το ίτερ. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο αντεπιχείρημα, ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες προσυπογράφουμε. Αλλά τώρα, δεδομένης ε, της ε, καταστροφής στην Επωνία και της διεθνούς κατάστασης, ίσως και άλλοι να είναι σε θέση να, πάρουν, να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε ολόκληρο το πρόγραμμα Ευρατόμ. Νομίζω ότι πρέπει να το επανασυζητήσουμε. Ίσως να μην αποτελεί τη βελτιστή λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, ταχύς ε, στις εναλλακτικέ. Ακόμη και το θέμα αυτό συζητείται και στη Γερμανία, ακόμη και από τους χριστιανοδημοκράτες, ότι πρέπει να είμαστε ε, ταχύτεροι στην επιτεύξη ενεργειακής αποδοτικότητα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να το λάβουμε πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα και να προσπαθήσουμε να έχουμε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέδια και project τα οποία είναι επικίνδυνα ε, και κοστίζουν σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι για να πρασινίσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, να μειώσουμε τις επιδοτήσεις ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. και να είμαστε έτοιμοι για τις μελλοντικές αλλαγές, ε, για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα. Αν θέλουμε να ε, πετύχουμε, να φτάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και τις κυβερνήσεις και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αιτιολογήσουμε ένα βαθμό ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και να έχουμε και παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη και ασφάλεια. Αν δούμε, παραδείγματο χάρη τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, το Εράσμου, τη διαβίωμα μάθηση, έχουμε πάρα πολύ καλή φιωρμογή, εξαιρετικά αποτελέσματα και πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν αυτά τα προγράμματα και υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να επενδύσουμε περισσότερο εκεί και αποτελεί τμήμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και νομίζω ότι πρέπει να αντικατοπτριστεί σε ε, στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο αυτούς τους τομείς. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, ε, θέλω να το τονίσω, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές ε, με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή να βασιζόμαστε μόνο στη Βουλή των Κρατών Μελών να δώσουν το 1% πάνω κάτω από το ΑΕΚΠΟΥΣ στο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα έχει ένα διαφορετικό σύστημα ίδιων πόρων και φυσικά ε, δεδομένης της κρίσης και των προβλημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή με την ακαμψία του προπολογισμού, η ευελιξία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Και εμεί ω πράσινοι είμαστε υπέρ του να γίνουν κάποιες αλλαγές, ε, ίσως να υπάρχει και κάποιο ειδικό περιθώριο αποθεματικού για ευελιξία εδώ και υποστηρίζουμε το να ε, έχουμε κονδύλια για τα αεφόρα προγράμματα υποδομών και θέλω να αναφερθώ και στο θέμα της διάρκειας. Στη δική μου ομάδα εξακολουθούν να, να λαμβάνουν χώρα συζητήσει ε, γιατί υπάρχουν ε, ε, πολύ καλά επιχειρήματα για 5, 7 και πάνω από 7 χρόνια. Αν ο προπολογισμό πρέπει να είναι πολύ χαμηλός, νομίζω ότι όπως πριν άλλη προηγμένως, είναι ρεαλιστικό το ζήτημα. Πρέπει να δούμε αν θα έχουμε διάρκεια 5 συν 5 και αν αυτό μας συμφέρει. Έτσι λοιπόν ε, είναι εδώ κάποια επιχειρήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε αλλά πρέπει να δούμε πώς έχει η σημερινή κατάσταση και ίσως να προσαρμοστούμε. Helga, jetzt. Ευχαριστώ Helga και τώρα ο Κόντρα Τσιμάνσκι. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem krytykę podniesioną tutaj w kilku wystąpieniach. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τις επικρίσεις που ακούστηκαν από τους ε, προλαλήσαντες και τις επισημάνσεις ότι θα πρέπει να δείξουμε πιο πολύ φιλοδοξία και παρησία στην έκθεση αυτή. Αλλά πρέπει να ζητήσουμε και ένα κοινό παρονομαστή. Έναν παρονομαστή που να εκφράζει και τις κοινέ μας θέσεις. Αυτός είναι ο τρόπος να εξασφαλίσουμε ώστε δυνατόν ευρύτερη υποστήριξη για τη θέση του Κοινοβουλίου από την Ολομέλεια και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στην έκθεση αυτό που βρίσκω θετικό είναι μεακές πτυχές. Ο εισηγητής με πολύ μεγάλη ε, σύνεση εφαρμόζει, χρησιμοποιεί όρους κλειδιά όπως κατάλληλη χρηματοδότηση. διατήρηση της υφιστάμενης χρηματοδότησης, η σπανίως αυξανόμενα ποσά, ενώ για τα γεωργικά, στις γεωργικές ε, πιστώσεις, αναφερόμαστε και σε μια πιο ε, κατανομή των πληρωμών. Πρέπει να είμαστε θέση να χρησιμοποιήσουμε τον όρο δίκαιη κατανομή των πληρωμών και σε αυτό επιμένω. Ωστόσο είναι λιγότερο ικανοποιητικό το κείμενο ως προς τις οριζόντιες πτυχές. Εδώ υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες και ασάφειες η έννοια του mainstreaming για διάφορες πολιτικές όπως την έρευνα, το περιβάλλον και το καθεξής, ε, την εισαγωγή δηλαδή των ενιών αυτών μέσα στις παραδοσιακές γραμμές του προϋπολογισμού. Ε, πώς θα γίνει αυτό όμως. Ε, εις βάρος των δαπανών που προβλέπονται για τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, Φερρυπίν Γεωργία. Και αν είναι έτσι, η περιβαλλοντική πολιτική σε ποιο βαθμό θα προσδιορίσει την έκταση των δαπανών για το Ταμείο Συνοχής, Φερρυπίν. Αυτό βέβαια είναι ένα δύσκολο ζήτημα, διότι θα πρέπει να ε, δείξουμε στον πολίτη τι θέλουμε, ότι έχουμε μια πολιτική συλλογή, συνοχής βεβαίως, ότι έχουμε μια γεωργική πολιτική βεβαίω, αλλά μπορεί ξαφνικά ο πολίτη, κοιτώντα αυτέ τι πολιτικέ να ανακαλύψει ότι υφίστανται νέοι στόχοι πλέον. Και αυτό δεν το βρίσκω σωστό. Αυτό μάλιστα το αποδίδω ως ε, συνέπεια στην ε, υπερβολική δίσδυση του κειμένου για το, 20, για το 2020 στην προσέγγιση αυτού του συγγετή. Είναι μάλλον ασαφές το κείμενο το σχετικό με την Ευρώπη 2020 και γι' αυτό θα προτιμούσα τον ε, προϋπολογισμό μας να τον εγγράψουμε μάλλον στα κείμενο των συνθήκων, να τον ευθυγραμμίσουμε προς το ρωστή στη διατάξη των ε, συνθήκων, γιατί εκεί είναι η πιο υγιής βάση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όχι συμπεράσματα που απαραίουν στη τελευταία ανάλυση από μία και μόνο σύνοδο κορυφής. Στους ιδίους πόρους. Η πεποίθηση ότι χρειάζεται να στηριζόμαστε περισσότερο στους ιδίους πόρους απορρέει από την πεποίθηση ότι έτσι θα αποφύγουμε την ε, αντιπαράθεση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ως προς την πρικοδότηση του προπολογισμού. Όμως, το να ανοίξει κατά την απόψή μου το θέμα των ιδίων πόρων αυτή τη στιγμή επιβαρύνει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει ή να επικεντρωθεί στην ε, διαμόρφωση ενός ποσού φορολόγησης ή στους φορολογικούς πόρους, και αυτό βέβαια έχει πολιτικό κόστος. Από τη μια μεριά δηλαδή εξετάζουμε το ενδεχόμενο να εξασφαλίσουμε πόρους από την ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά ταυτόχρονα με αυτό επιβαρυνόμαστε με διπλή, διπλό πρόστιμο, γιατί τα ποσά του ETS που θα έπρεπε να επενδύονται στα κράτη-μέλη αντί να πάρει σε αυτό το σκοπό, αντί να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση δηλαδή, επιστρέφουν στις Βρυξέλλες για να δαπανηθούν σε αυτό το επίπεδο κατά τρόπο αυθαίρετο. Αυτό είναι αντίθετο με τη συμφωνία για το ETS. Επίσης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, και αυτή είναι τελευταία μου παρατήρηση, πολύ μεγάλη εξειδίκευση για να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι σύμφωνη με τις, ε, με τις εξελίξεις στην παγκοσμιοποίηση η φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Φορολογίας την φορολόγηση των επιχειρήσεων, έχουμε κλείσει το μέλλον της Ευρώπης ανεξαρτήτων στόχων, ανεξαρτήτων στόχων και προτεραιοτήτων. Κυρία Χάουκ, μια παρατήρηση αν μου επιτρέπετε. Σας παρακαλώ αν θέλετε κάπως να συνοψίζεται, διότι στην έκθεση που θα προκύψει από την Επιτροπή μας δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για φόρο. Όποιος και είναι αυτός. Θα πρέπει να το αποφύγουμε. και να το σημειώσουμε αυτό και στην έκθεση του Σαλβαδόρου, ότι θέλουμε, εάν υπάρξει φόρο, όποιο φόρο είναι αυτό, εμεί θέλουμε μόνο να σημειώσουμε τι είδου χρήση θα έχει, τι είδου λειτουργία θα έχει. Δεν υπαγορεύουμε όμω τι είδου φόρο θα πρέπει να εισαχθεί γιατί και δύσκολο θα είναι να συμφωνήσουμε εμεί, αλλά και ταυτόχρονα θα αποτελούσε ένα κίνδυνο αυτό να παραβλέψουμε κάποιε περαιτέρω ε, συνέπειες περιπλοκέ που θα μπορούσε να έχει η εισαγωγή ενό τέτοιου φόρου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για φόρο. Ούτε για το δεξίδιο του άνθρακα, ούτε για τι επιχειρήσει ούτε για τίποτα. Μόνο θα πούμε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει εισαγωγή ενός νέου φόρου, θα πρέπει αυτός να ικανοποιεί αυτούς και αυτούς τους στόχους ή τις προϋποθέσεις καλύτερα. Αυτό για να μην παρασυρθούμε σε τέτοια συζήτηση. Παρακαλώ κύριο Σπόρτος. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Θα εκφράσω μια προσωπική γνώμη γιατί στη δική μου ομάδα σίγουρα θα υπάρχουν και προσεγγίσεις επισημαντικών σημαντικών ε, που είναι διαφορετικές. Ε, αλλά εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω από αυτή την προβληματική των πόρων. Αναπόφευκτα πρέπει να ξεκινήσω από αυτό, γιατί νομίζω ότι όταν μιλάμε για δημοσιονομικές προοπτικές, από το 2014 και μετά βρισκόμαστε στα έναν ορίζοντα όπου τα στρατηγικά προβλήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος θα τεθούν αναπόφευκτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δυνατό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα σταθερό νόμισμα, το ευρώ, δίχως να έχει και σταθερό προπολογισμό. Και αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικό, ουσιαστικό για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση γι' αυτό μέσω του προπολογισμού. Πρέπει να οικοδομήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο Ταμείο σταθερότητα και να έχουμε μια στρατηγική για την χορήγηση κονδυλίων, για τα μεγάλα project και για άλλα είδη προγραμμάτων. Αυτή η στρατηγική που είναι κατακαιρματισμένη δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν το πρώτο που θέλω να πω είναι ακριβώς αυτή η επιλογή. Τώρα, δεύτερη πτυχή αυτής της πρώτης εκτίμησης εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ένα παγιωμένο προϋπολογισμό ανεξάρτητα από, τον ακριβή, από το ακριβές του μέγεθος, διατηρώντας την αρχή που τον έχει ε, που τον διέπει μέχρι σήμερα, δηλαδή η χρηματοδότηση μέσα από τα κράτη-μέλη, για έναν απλό λόγο. Γιατί όλα τα κράτη έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή να δίνουν όσο δυνατόν λιγότερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να λαμβάνουν όσο δυνατόν περισσότερα. Και έτσι λοιπόν βλέπετε ότι εδώ διακυβεύονται πολλά και θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Ένα τρίτο πρόβλημα που πρέπει να εξετάσουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δώσει μία υπόσχεση κοινωνικής σύγκλησης. Δηλαδή αυτό που μας έδειξε αυτή η κρίση ήταν ότι οι πολιτικές συνοχής δεν αρκούν. Είναι ανεπαρκείς για να εγγυηθούν μια στρατηγική κοινωνική σύγκληση. Εμείς σε επίπεδο κάθε χώρας μπορούμε να αποφύγουμε την επιδείνωση των ενισοτήτων. Αλλά δεν κατορθώσαμε να αποφύγουμε την επιδείνωση αυτή των ενισοτήτων ε, μεταξύ χωρών με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Εγώ βλέπω τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ως ένα εργαλείο καταπολέμησης των αποκλήσεων, που είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Λεχθέντως αυτού. Πιστεύω ότι η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά θετικών στοιχείων επί των οποίων πρέπει να εργαστούμε για να καταλήξουμε σε διευρυμένη συνένεση. Όμως είναι μία έκθεση που δεν τολμά ιδιαίτερα και υπάρχουν και αντιφάσεις. Δεν ε, μπορούμε να αποδίδουμε φιλοδοξίες στο προϋπολογισμό της φιλοδοξίας που αποδίδει αυτή η έκθεση με μια πρόταση προϋπολογισμού η οποία συνοψίζεται στο 1,23% του Ευρωπαϊκού ΕΚΠ. Και προφανώς είναι μια δυσαναλογία αυτή μεταξύ, υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των πόρων και των φιλοδοξιών. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι εμεί στην Ευρώπη δεν έχουμε μία στρατηγική για την ανάπτυξη η οποία να δημιουργεί ε, αϊφόρους μηχανισμούς προσφοράς. Για μένα το κύριο πρόβλημα της ανάπτυξης και της σύγκλησης είναι αυτό των πολιτικών που σταθεροποιούν την ζήτηση. Αυτή είναι μια διαφωνία που έχω λοιπόν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι ίσως και το κύριο παράδειγμα. Ε, σωστά επενδύουμε στην ε, εκπαίδευση, στην διαβίου μάθηση και στην έρευνα, αλλά δεν είναι συνεπές να καταδικάζουμε όλες τις νέες γενιές στην επισφάλεια ε, στην ε, ανάπτυξη και στην έρευνα, στην αγορά εργασίας ε, που κατόπιν προέρχεται από την έλλειψη, παραδείγματος χάρη στη διαβίου Αυτή η πτυχή δεν υπάρχει καθόλου στην έκθεση του συναδέλφου. Ευχαριστώ, Μιγγέλ. Αν σωστή ήταν η μετάφραση, γιατί δεν καταλαβαίνω τα πορτογαλικά από το πρωτότυπο. Αν ήταν καλή η μετάφραση, μίλησες και είπες ότι μόνο 1,23 ε, ΑΕΠ θα δώσουμε. Μα τι να σας πω, μακάρι, μακάρι να το πετυχαίναμε αυτό, το 1,23%. Κύριε Φοντάνα, είστε εσείς ο εκπρόσωπος ε, του EFD. Όχι. Α, δεν έχουμε λοιπόν ε, κανέναν εδώ πέρα. Άρα να δώσω το λόγο στον Ράινερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σχέδιο έκθεση του Σαλμαδόρ συνολικά είναι πάρα πολύ ισορροπημένο και περιλαμβάνει πάρα πολλά καλά στοιχεία και αποτυπώνει αυτά που είχαμε συζητήσει από κοινού. Και θα έχουμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε και στο εσωτερικό των ομάδων και μεταξύ των ομάδων το συνολικό πακέτο. Και φυσικά τώρα ξεκινάει και η μεγάλη πίεση από τη δημόσια γνώμη και θα πρέπει να, να προσέξουμε να μην ε, καταλήξουμε σε μια συνάθρηση μεμονωμένων ε, συμφερόντων. Να πω το εξή, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως, αυτά τα συντηρητικά στοιχεία του προϋπολογισμού εγώ θα πρέπει να μιλήσω και να πω το αντίθετο, γιατί το συντηρητικό στοιχείο του προϋπολογισμού σημαίνει και μία συνέχεια. Νομίζω ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φύγαμε το, τη γενιά των χρεών ή τις επόμενες γενιές. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ενιαίο σχέδιο και να υπάρξει επικέντρωση όχι μόνο στο 1% αλλά και στο 23% ή οποιοδήποτε ποσοστό, αλλά να δούμε συνολικά την πολιτική προϋπολογισμού, τη δημοσιονομική, να δούμε συνολικά τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τι θα πρέπει να πετύχουν στην, στο πνεύμα του ευρωπαϊκού project. Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ιστορικό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Επί 15-20 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεράσπιζε μόνο τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την τελευταία φορά εξετάσαμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθήσαμε να δώσουμε μεμονωμένε εμφάσει από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και τώρα το Κοινοβούλιο ε, για πρώτη φορά πριν καταθέσει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τέτοια θέματα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και προαπαιτεί και μεγάλη προσπάθεια ε, από εμάς. Και επίση ε, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η διεθνής πραγματικότητα και αυτό φυσικά επηρεάζει και τις προτεραιότητές μας και Φυσικά χρειάζονται και τα απαραίτητα αποθεματικά και η απαραίτητη ευελιξία στον προϋπολογισμό προκειμένου στο συντορικό ενός ε, δημοσιονομικού πλαισίου είτε είναι πενταετές, δεκαετές ή επταετές, να έχουμε πάντα τη δυνατότητα και πάντα δεν υπάρχει δυνατότητα ε, αν υπάρχει σωστή διαχείριση δια... που δεν υπάρχει ακόμα σήμερα αν υπάρχουν ε, οι προϋποθέσεις αυτές, ε, να συζητήσουμε το πενταετές πλαίσιο, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που είναι καθοριστικό δε είναι, και αυτό είναι μέρος του όλου οράματος Γκέραν, να κοιτάξουμε τον διακυβερνητικό χαρακτήρα και να μην επιτρέψουμε να υπονομεύσει τον κοινωτικό χαρακτήρα. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τους κινδύνους και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα ειδικό κεφάλαιο για το τι περιλαμβάνεται σήμερα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, τι διοργανώνεται σε διεθνές επίπεδο και τι ποσά εμπλέκονται. Είναι πραγματικά τεράστια. Νομίζω ότι έτσι θα, καταδείξουμε και στην, θα καταδείξουμε και στην κοινή γνώμη ότι κοιτάξτε αυτά είναι τα πράγματα με τα οποία θα συμφωνούμε. Θέματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας προκειμένου να κοιτάξουμε τις διάφορες διαστάσεις. Να πω το εξή. Φυσικά, σε κάθε ε, στήλη και κεφαλίδα του προπολογισμού μπορεί να γίνουν ε, αποταμιεύσει. Και δεν είμαστε ειλικρινεί άμα δεν το προτεχτούμε αυτό. Και αν δεν μιλήσουμε για αρνητικέ προτεραιότητε, θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να κάνουμε μία ε, περικοπή σε όλες τις γραμμές και μετά να κάνουμε συζητήσεις και να δούμε ποιος ε, μπορεί να αποδείξει ότι χρειάζεται να επανέλθουν ε, τα ποσά αυτά σε κάποια συγκεκριμένη ε, γραμμή και να πούμε λοιπόν στο Συμβούλιο τι κάνετε με τις διαρκείς σας δεσμεύσεις 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη. Μα τι να κάνουμε αφού μας λείπουν 120 σε κάθε χρόνο υποχρεωνόμαστε να δίνουμε 0,7 σε αναπτυξιακή βοήθεια και το ποσοστό αυτό είναι 0,4%. Τι σημαίνει αυτό, 30 ε, εκατομμύρια επιπλέον. Μα τι θα πρέπει να πούμε, να πούμε ότι δεν είναι εφικτό, με πάσα ειλικρίνεια, ή να το αφαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη. Νομίζω επίσης ότι το θέμα είναι να συζητήσουμε ασφαλώς το πώς θα διατηρηθούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συζητήσουμε πώς θα τα προασπίσουμε. Στη διαδικασία θα ήθελα να παρακαλέσω να θέσουμε την συνεργασία ακόμα πιο πολύ στο επίκεντρο και να απειλήσουμε ότι αν δεν συνομιλήσουν μαζί μας μπορεί να αναγκαστούμε να πούμε όχι. Αυτό από πλευράς διαδικασίας και για τα ίδια μέσα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. Ακούσαμε όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Έχω τώρα τις επιμέρους παρεμβάσεις και ένα χρονικό περιθώριο περί τα δύο λεπτά για τον καθέναν. Μπράντι, Σποκόφσκ, Χρυπνά. Λεφόλ. Άλλος θέλει το λόγο. Μάνσος, να σας σημειώσω. Κοτμάνης. Σκέσκι. Μάλιστα, Ιούγκ. Hm. Ίσα ίσα θα τα προλάβουμε. Δύο λεπτά ο καθένας. Για να συνεχίσουμε μετά. Δεν θα σχολιάσω εγώ γιατί συνήθως κατηγορούμε το Συμβούλιο γι' αυτά. Δεν ε, θα ήθελα να πέσω αυτή την παγίδα τώρα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Γαρίγα για την έκθεση του. Αποτελεί μια πολύ καλή ε, έκφραση των όσων έχουμε συζητήσει, χωρίς βέβαια να αποτελεί και την λύση για τον τεράστιο γόρδιο δεσμό που έχει πάνω στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων η Ευρώπη και ας είμαστε ρεαλιστικές, ρεαλιστές, έχουμε ένα τεράστιο γόρδιο δεσμό, περίπλοκο. Διαφορετικά συμφέροντα των διαφορών κρατών μελών. Έχουμε εκείνα που εισφέρουν στον προπολογισμό που θέλουν να παγώσουν. Θέλουν εκείνα που, ε, υπάρχουν εκείνα τα οποία θέλουν να πάρουν περισσότερα γιατί εισπράττουν από τον προπολογισμό. Έχουμε τα καινούργια κράτη-μέλη που επιτέλους θέλουν να συμμετάσχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και όλα αυτά βέβαια τα αντικρουόμενα συμφέροντα και αιτήματα δεν είναι εύκολο να συγκεραστούν. Είμαι πεπισμένο πάντως ότι η μόνη λύση είναι να κοιτάξουμε με σοβαρότητα, να αναζητήσουμε δημιουργικές εφάνταστες λύσεις και να μην περιοριστούμε μόνο σε έναν απλό προϋπολογισμό, αλλά να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε στους διάφορους τομείς ε, και στους διά, στις διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού τα κονδύλια. Γιατί μέχρι στιγμής κάνουμε μόνο αυτό, κοιτάμε τον προϋπολογισμό δηλαδή. Και γι' αυτό θα παρακαλέσω να μην ε, κάνουμε εμεί οι ευρωβουλευτέ την ίδια δουλειά που κάνουν τα κράτη-μέλη, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε μόνο ή να επιδιώξουμε να εξυπηρετήσουμε μόνο τα εθνικά συμφέροντα. Να στοχεύσουμε περισσότερο στο ευρωπαϊκό συμφέρον εμεί. Και θα ήθελα να επενθυμίσω, το 2005 προσδιορίστηκαν οι δημοσιονομικέ προοπτικές επί Προεδρία Τόνι στο Συμβούλιο και αυτό που πράττουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε λίγο πολύ το πώς θα ε, λειτουργήσει ο προπολογισμό, τι κονδύλια θα δαπανούν μέχρι το 2020. Ε, είμαστε λοιπόν πιο ε, φιλόδοξες, έχουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα. Τώρα η Κίνα ξέρετε ότι έχει καταθέσει το πρόγραμμά τη όχι μόνο μέχρι το 2015 και το 20, αλλά πιο πέρα από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμεί να κοιτάξουμε και την καινοτομία και την δημιουργία. Όχι μόνο τα χρήματα που θα βάλουμε δηλαδή στα προγράμματα αυτά, αλλά το πώ θα λειτουργήσουμε τα, τα προγράμματα αυτά, πώ θα δαπανίσουμε τα κονδύλια που δαπανούμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω καταρχήν ευχαριστώντας ε, τον Σαλβαδόρ. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι το έγγραφο πραγματικά αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας. Όμως ε, υπάρχουν πολλά αλλά. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καθώς ε, δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να σου ζητήσω, Σαλβαδόρ, να σκεφτείς ε, μια αναδιάρθρωση του πίνακα που έχει στη σελίδα 18 γιατί αυτή η κατηγοριοποίηση δεν αντικατοπτρίζει πολύ καλά ούτε καν τις δικές σου προτεραιότητες, πόσο μάλλον των υπολείπων η κατηγοροποίηση θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει και θετικές και αρνητικές προτεραιότητες και δεν νομίζω ότι αυτοί οι υποτομείς θα πρέπει να παραμείνουν ε, ως έχουν, γιατί αυτοί είναι πιο σημαντικοί από τους ίδιους τους τομείς. Από τους ίδιους φακέλους, αν θέλεις να, δει, να δεις ε, ε ανάπτυξη ε, και δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτό είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να γίνει μια διάφραση σε σχέση με του τομεί. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό το πώ θα έχει παρουσιάσει εδώ και αν θέλουμε πραγματικά προτεραιότητες, ε, ίσως ε, θα έπρεπε να τις βάλουμε όλες στο πρώτο τομέα και να δούμε αν μπορούμε να δαπανίσουμε περισσότερα από αυτόν και να δούμε τι σημαίνει για το δεύτερο τομέα και τα υπόλοιπα. Τώρα, για τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει πιο ψηλά στην ιεραρχία, γιατί θα μας κοστίσει πολλά. Κυρίως ε, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή και ο μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Για να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά και μοιάζεται παντός. Είμαστε μόνο σε μια πρώτη φάση, συζητούμε γενικά. Αυτό που τώρα λέω νομίζω ότι θα πήγαινε περισσότερο στη συζήτηση του απογεύματο, όπω την έχουμε προβλέψει, αλλά εν Ο επόμενο ομιλητή. Η ομιλήτρια. Ντανούτα Χιούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη δουλειά του Σαλβαδόρ, τι προσπάθειέ του, τι δικέ του και των συναδέλφων του και θα ήθελα να επισημάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η ε, απευθείας χρήση του Ευρωπαϊκού προβολισμού δεν αποτελεί την τελική λύση στην, ε, στις μεγάλες προκλήσεις της δημοσιονομικής που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για τη σημασία που ναι, αποδίδεται στον καταλητικό και μοχλευτικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό περισσότερο για το συντονισμό των, ε, της χρηματοδότησης επί Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένους τομείς πολιτικής που θα έχουν και ζωτική σημασία ή θεμελιώδη καλύτερα σημασία για το μέλλον μας. Και πάνω απ' όλα ε, συνδυασμό χρηματοδότησης για τον οποίο νομίζω πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση μεθοδολογία ή μια διευκόλυνση, ένα μέσο διευκόλυνση που θα επέτρεπε το συντονισμό τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το δεύτερο σχόλιο. ακούω συναδέλφου να λένε δεν υπάρχει αλλαγή, βλέπουμε όλε τι ίδιε πολιτικέ και τον ίδιο προπολογισμό. Σε αυτού του συναδέλφου θέλω να απαντήσω ότι δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε πιο προσεκτικά τι πολιτικέ. Οι περισσότερε ευρωπαϊκέ πολιτικέ έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια μέσα από μια διαδικασία θέτει των μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο τη κρίση και εν ώψη τη προετοιμασία για την Ευρώπη 2020. Και παρακαλώ, τους συναδέλφους που επισημαίνουν τέτοιου είδου ε, ομοιότητα με τους προηγούμενους προπολογισμού να αντιληφθούν ότι δεν πρόκειται για ε, τις ίδιες πολιτικές και την ίδια αξιοποίηση. Για την έρευνα και ανάπτυξη. μίλης λησμονείτε παρακαλώ ότι έχουμε κατά 159% ενισχύσει τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό Πολιτικό. 159% για τον Ευρωπαϊκό υπολογισμό. Όταν λένε οι συνάδελφοι ότι πρέπει να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε τι δαπάνε, κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά ποια είναι η χρηματοδότηση τη τώρα. Εκεί που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση θα είναι το πώ θα αξιοποιούνται τα κονδύλια και πώ θα είναι πιο αποτελεσματική αυτή η αύξηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί. Και επίση θα πρέπει να προσδοριστούν πιο, σαφεί όροι για τη συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και βέβαια να αλλάξει και ο τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια μα. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό επίση. Στο 121 σημείο του Σαλβαδόρου, συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, ε, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, που είναι ένα σημείο το οποίο θεωρώ ζωτική σημασία. Και θα πρέπει να καλέσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρουν μια λύση, ε, μια μέθοδο εργασία και συνεργασία για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει διαρκώ ή να συμμετέχει διαρκώ στι διαπραγματεύσει αυτέ. Ευχαριστώ, Στεφάνο. Θέλω να χαιρετήσω το έργο που μας παρουσιάστηκε και την γενική ισορροπία που διαπιδοκείμενο Τώρα στους στόχους που προσπαθεί να επιδιώξει και που εγγράφονται στην ε, περιβόητη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στις προτάσεις οργάνωσης ε, του μελλοντικού προπολογισμού με τις διάφορες συνιστώσεις ε, για την εφορία ε, την ανάπτυξη, την ηθαγένεια, την ε, χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση κτλ. Κοιτάξτε, προσοχή να μην ε, συνοψίσουμε τις μεγάλες πολιτικές, την ΚΑΠ, την κοινήλευτική πολιτική κτλ. Να μην τις παρουσιάσουμε με ένα συνοπτικό τρόπο, γιατί υπάρχει ένας οικονομικός τομέας που κρύβεται πίσω από αυτές τις πολιτικές. Όμως θα ήθελα να στραφώ στο θέμα των ιδιών πόρων. Όλοι έχουν κάποιες ιδέες ε, για το ποιες θα μπορούσε, ποιοι θα μπορούσαν να είναι ήδη οι πόροι στο μέλλον για την Ευρώπη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες. Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε πρόσφατα σε μία έκθεση υπέρ ενός πόρου για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όμως ε, δεν μου φαίνεται να αρκεί η ιδέα που αναφέρεται στο 118 για την ε, δυνατότητα ε, να υπάρχουν ήδη πόροι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη σαφήνεια να φέρουμε τη φιλοδοξία που έχουμε να έχουμε ίδιους πόρους, όχι ενδεχομένως και αυτή είναι η συζήτηση που θα έχουμε για το θέμα της συνοχής, της δομής, της σχέσης μεταξύ εσόδων, εξόδων, στόχων. Πραγματική μάχη για το Κοινοβούλιο, για να λάβουμε υπόψη ε, την Ευρωπαϊκή Διάσταση και να βγούμε από το διάλογο που γίνεται μεταξύ των κρατών για τον προπολογισμό όπως γίνεται σήμερα, είναι να έχουμε ίδιους πόρους και αυτό πρέπει να το λέμε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δύο λεπτά δεν μου φτάνουν. Πιστεύω ότι το πιο θετικό από αυτά που διάβασα ήταν αυτή η μόχλευση. Αυτή η μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό είναι το βασικό. Το PPP δεν... Ε, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν ε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο πώς μπορεί να εμβαθύνουμε στις ε, συμπράξεις αυτές. Γιατί καταρχάς υπερισχύ, μάλλον κανονικά το, τα, οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι υπαριθμόν ένα. Και το θέμα είναι και το πώς θα το γράψουμε αυτό, γιατί διαφωνώ λίγο με τον, με τον κύριο Καρίγκα Θεωρώ ότι ο συντονισμό μεταξύ των επιτρόπων είναι αυτό που εννοούμε εις βάθος. Κοιτώντας τον υπολογισμό βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά κονδύλια τα οποία δεν ταπανώνται σε διάφορους τομείς που μάλιστα επικαλύπτονται με άλλους τομείς. Για παράδειγμα, για τα προγράμματα ε, ε, επιστήμης, για παράδειγμα, για προγράμματα ε, γεωργίας και βλέπουμε ότι δεν ταπανώνται. Ο συντονισμός, για παράδειγμα, μεταξύ της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου στην γεωργία και των διευθυντικών ταμείων είναι τεράστια καταστροφή παίρνουμε ένα εκατομμύριο από τον ένα κλάδο και τον παίρνουμε στον άλλο κλάδο. Και η πρόσθετη αξία είναι ότι ο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων ε, επιτρόπων, που είναι ο καθένα ε, αρμόδιος για διαφορετικούς επίπεδους, θα πρέπει να γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται εδώ ένα επίτροπο και να λέει ότι δεν έχω χρήματα. Να το ρωτάμε, μα πώ συνεργάζεται με τον άλλο επίτροπο και να μα λέει Α, θα αρχίσουμε συζητήσει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί μια βάση για τι μετέπειτα ε, ε, διαπραγματεύσει μα. Η πρόεδρο. Νομίζω ότι, ότι το τελευταίο αυτό που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι επίτροποι θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Γιατί για παράδειγμα, το έχουν σκεφτεί μάλλον η Επιτροπή αυτό, γιατί έχουν στείλει σχετικέ επιστολέ που αναφέρουν τι κοινέ αυτέ ε, συζητήσει. Τώρα, κατά πόσο θα ακολουθήσουν αυτά, θα δούμε. Ο κ. Σικεύσκη. θέλει συγκέντρωση το όνομά σας. Ευχαριστώ για να αναδιατυπωθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύσκολο διατηρώντας θέματα βιωσιμότητας. Θα πρέπει να βρούμε και να τηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των αλλαγών που θέλουμε και των, της συνέχειας που θέλουμε να υπάρχει προκειμένου να μην καταστούν ε, πολύ εξικέλευτες αυτές οι αλλαγές. Είναι πολύ ισορροπημένη η πρότασή σας. Αλλά αναγκαζόμαστε εδώ πέρα να περιορίσουμε τα δημοσιονομικά μας μέσα. Αυτό επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητάνε πάντα από τους ε, βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου να αναπτύξουν ε, μια, ε, ένα όραμα σχετικά με τα θέματα αυτά και εδώ πέρα τονίζονται η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα κυρίως. Αυτές οι δύο πτυχές, η ανάπτυξη φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ανταγωνιστικότητα δεν ε, προωθείται και ενισχύεται μόνο μέσω κονδυλίων, αλλά και μέσω διευκόλυνσης των σχετικών όρων. Η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται με τη μείωση των ε, επιβαρύνσεων για τις εταιρείε. Και αυτό φυσικά συνεπάγεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης τα τελευταία 20 χρόνια. Πληρώσαμε τον περιορισμό της παραγωγής της γεωργίας. Και πάντα αναφέρουμε και μιλάμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Είναι όμως ε, σημαντικό η γεωργία, η ΚΑΠ να διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο, γιατί εδώ πέρα τίθενται και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Η Κορνέλη Στεγιόμ. Και μετά το λόγο έχει ο Σαλβαδόρ και πάλι. Ο κύριος Στεγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ρωτήσατε θέματα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην, ε, στο Ζέλαντ, ε, στην ε, Ολλανδία, η χρηματοδότηση είναι δύσκολη και γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε όραμα. Είναι πολύ δύσκολη η χρονική συγκυρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει σαφείς επιλογές, δεν έχει κάνει σαφείς επιλογές εδώ πέρα στην έκθεση. Στα ταμεία θα έπρεπε να πούμε ότι το να αντλούμε χρήματα από την Ολλανδία, από μικρά project τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά, τα οποία δεν βελτιώνουν την Ευρώπη. Αυτό που θέλουμε είναι συγκέντρωση των ε, κονδυλίων, για παράδειγμα, για θέματα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ε, μεταρρύθμισης ε, της γεωργικής πολιτικής και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων. Αν το τορμήσουμε αυτό, αν κάνουμε σαφείς επιλογές. Αν επικεντρωθούμε με τους δαπάνες, με τους πόρους, σε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, εκεί σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να βγάλουμε κέρδος. Τα μικρά προγράμματα να τα αφήσουμε κατά μέρος. Ένα παράδειγμα άλλο να σας δώσω. Μιλήσαμε στην Επιτροπή ενία Ενίας αγορά Αγοράς για τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προγράμματα για τον τουρισμό στην Ευρώπη, τα οποία δεν βελτιώνουν, θεωρώ, ιδιαίτερα την Ευρώπη. Να επικεντρωθούμε λοιπόν, να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες για να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια εποχή λιτότητας, όχι να γράφουμε μια έκθεση όπου ουσιαστικά συμπεριλαμβάνουμε τα πάντα και πάλι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο Σαλβαδόρ. Eh. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι όταν ε, κάνω συνόψεις ε, δεν ε, απαντώ συνήθως, όμως τώρα θα αναφερθώ γενικά στα σχόλια που ακούστηκαν και κατόπιν στη διάρκεια της συζήτησης θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και στη διαφορά με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές που αντιδρούσαμε σε προηγούμενη πρόταση, σήμερα η προηγούμενη πρόταση είναι δική μας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ προσπάθησα λοιπόν να υποβάλω μια πρόταση όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη και γνωρίζω φυσικά ότι όλοι εσείς ε, έχετε τις δικές σας προτεραιότητες ε, και φυσικά ξέρετε ε, ότι εδώ πολλές φορές πυροβολούν τον πιανίστα. Οι υπόλοιποι όμως εγώ προσπάθησα εδώ να συνθέσω τη μουσική που όλοι ε, επιθυμείτε και με ουστάρισα σε όλους σας. Πάντως σας ευχαριστώ για την κριτική σας. Ε, άκουσα τον άλλο που είπε ότι ε, έχουμε συντηρητική προσέγγιση. Κοιτάξτε, είναι συντηρητική αυτή η προσέγγιση και δεν έχει διάφορες κομματικές αποχρώσεις γιατί το θέμα έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Εδώ ε, κοιτάξτε, αν δούμε πώ πήγαν αυτέ οι δημοσιονομικέ προοπτικέ, δεν πήγαν και τόσο άσχημα. Μπορέσαμε να πετύχουμε πολλού από του στόχου. Υπάρχουν πολλέ ελλείψει, αλλά εγώ νομίζω ότι η βάση αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών είναι καλή και πρέπει να αποτελέσει και το δρόμο για τι επόμενε. Τώρα, ε, αν είναι επικίνδυνο ή όχι, εγώ νομίζω ότι η δομή που προτείνουμε ενέχει ένα βαθμό κινδύνου, δηλαδή ε, βλέπουμε και σήμερα στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές υπάρχει ένας βαθμός κινδύνου. Ε, δεν... Ε, ε, ε δεν ακολουθούμε εδώ τι επιθυμεί κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κάποιο εθνικό κοινοβούλιο. Εδώ ακολουθούμε τις ε, προτεραιότητες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε σε πιο δύσκολη θέση όπω καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να προσπίσουμε και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και είναι πιο δύσκολο ο ρόλο μα τώρα για τη λιτότητα. Νομίζω ότι ε, πρέπει εδώ να δούμε ποιε εξοικονομήσει μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρετε πώ έχει η κατάσταση. Τώρα, να σας πω ότι εμείς ε, πρέπει να δείξουμε ότι είναι αδύνατο να ξοδέψουμε ε, λιγότερα, αλλά και ταυτόχρονα δεν μπορούμε ούτε περισσότερα να δαπανίσουμε. Πρέπει να ξεβρούμε μια δημοσιονομική ισορροπία για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Τώρα, αυτές οι αποτομιεύσεις θα γίνουν μέσω των αρνητικών ε, προτεραιοτήτων. Ε, κοιτάξτε, σε αυτές τις εκθέσεις της μεσοπρόθεσμες που παρουσιάζονται για τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα ειλικρινά δεν είδα σε καμία περίπτωση αρνητικές ε, προτεραιότητες όλες ε, είναι αισιόδοξε και μάλιστα σημειώνω ότι μπορούν να βελτιωθούν και τα προγράμματα όμως υπάρχουν σε αυτές τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις ε, συστάσεις αν υπάρχουν μάλλον τέτοιες συστάσεις για αρνητικές προτεραιότητες εγώ δεν τις είδα η μόνη αρνητική προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε εμείς ε, είναι ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τις δαπάνες ε, για την Αλφού Τρούπε. Ε, κοιτάξτε, αναφέρεται φυσικά η ενεργειακή αποδοτικότητα στο εσωτερικό των πολιτικών προκλήσεων και των προτεραιοτήτων και για την κοινή αγροτική πολιτική φυσικά θα είναι πιο πράσινη. Εμείς δεχόμαστε την μεταρρύθμιση που προτείνει ο Επίτροπος Όλος ε, χωρίς να μειώσουμε τις επιδοτήσεις αλλά φυσικά όσο περισσότερο πιο φιλική προς το περιβάλλον αυτή η πολιτική, τόσο περισσότερο συμφωνούμε. Κοιτάξτε, τώρα κύριε Ζημάσκη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για το ποιος πληρώνει ποια πολιτική. Ε, πρέπει εμείς να απαντήσουμε σε μια ανακατάσταση, επομένως θα υπάρχουν και νέες προτεραιότητες, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάρος των πολιτών που είναι σε πιο ευάλωτη θέση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύω εγώ, γι' αυτό διατηρώ μέσα στη δομή την πολιτική συνοχής ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους υποτομείς της στρατηγικής το 2020. Θέλω να επισημάνω ότι συνεχίζει να είναι σημαντική η πολιτική συνοχή τώρα για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων. Αν θα έχει πολιτικό κόστο. φυσικά. Φυσικά και θα έχει. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων αυτό που δεν πρέπει να έχει είναι κόστο για τον πολίτη. Κόστος για τους πολιτικούς, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κόστος για τους φορολογουμένους. Γι' αυτό προτείνουμε ουδέτερη πολιτική εδώ. Το ίδιο και για το συνάδελφο Πόρτα. Η στρατηγική για το 2020 ακριβώ έχει μία συνιστόσα κοινωνική. Ο έσχατο στόχο τη στρατηγική αυτή είναι η δημιουργία θέσεων εργασία μέσω τη ενίσχυση των ε, διάφορων ειδών ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία καλύτερη κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή που δημιουργεί θέσει εργασία. Δέχεται οποιαδήποτε πρόταση μέσω τροπολογιών, είμαι ανοιχτό. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε τι θα γινόταν με τις χώρες που σήμερα είναι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής αν ε, δεν υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η σημαντική προσπάθεια ε, η μεταφορά πόρων από τις πιο πλούσιες στις λιγότερο πλούσιες χώρες, ε, χωρίς την πολιτική συνοχής, θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη σήμερα στην Βέγε. Εγώ κατοπτρίζω εδώ τις συζητήσεις και απλώς θέτω ένα κοινό παρανομαστή ίσως να είναι λιγότερο φιλόδοξο όλα αυτά από το να προσπαθήσουμε να καταγράφουμε εδώ μία καινοτόμο θέση. Όμως, όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να, διατη, να τουλάχιστον 500 ψήφους στην Ολομέλεια για να προσφέρουμε μία καλή πολιτική πρόταση με τον προπολογισμό δεν γίνεται επανάσταση, κυρίω όταν εξαρτώμαστε από 27 υπουργού οικονομικών και εθνική οικονομίας ε, και είναι σε απελπισμένη κατάσταση ε, τα δημόσια οικονομικά του στη χώρα του. Έτσι λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα και όταν θέτουμε έναν προπολογισμό που έρχεται ως συνέχεια ε, εδώ Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και φυσικά προβαίνουμε και σε ένα εγχείρημα που πολιτικά να είναι παρακινδυνευμένο. Γι' αυτό τα έχω παρουσιάσει έτσι στην έκθεση αυτή και φυσικά εμείς σεβόμαστε ότι είπαμε πάντα στην Επιτροπή Προπολογισμού για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών χρειάζονται νέοι πόροι, νέα χρήματα. Αυτό υπάρχει και συνεχίζουμε να το θέτουμε στην έκθεση εγώ αναλύω τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις ε, και συνάγω ότι φυσικά χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση. Τώρα πώ θα επιτευχθεί αυτή η χρηματοδότηση βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα μιας πολιτικής δήλωση. Δεν ξέρω αν εσείς τελικά μετά από τη συζήτηση των τροπολογιών που θα έχετε προτείνει θα προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις, όμως είναι και εντολή τη Επιτροπής ΣΟΥΡ να αποδείξει ότι πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση, γιατί δεν επαρκούν οι σημερινοί πόροι για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είμαι στη διάθεσή σας ε, να αναθεωρήσω και τη δομή του κειμένου, πάντα μπορεί να βελτιωθεί, αλλά θέλω να σας πω ότι ε, ο στόχος είναι ο εξής, να είναι όσο δυνατόν πιο ορατή, να προβληθεί όσο δυνατόν περισσότερο στρατηγική για το 2020, γιατί έχει ψηφιστεί από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο και θα ψηφίσετε πιθανότητα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι θέλουμε να πετύχουμε περισσότερε θέσει τα επόμενα χρόνια. Θέλω να το καταστήσω αυτό ορατό, να το προβάλλω και θέλω όλε τι πολιτικέ να τι συμπεριλάβω σε αυτή τη δομή. Κοιτάξτε, ας ε, θυμόμαστε ότι τελικά εδώ μιλάμε για μια πολιτική δήλωση. Ας προσπαθήσουμε να είναι στο δυνατόν ε, πιο ευανάγνωστη η δήλωση αυτή και να λάβει το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή. Βέβαια, αν ε, είναι δυνατό, θα βελτιώσουμε ορισμένα σημεία. Όμω, εγώ θέλω να τονίσω την έλλειψη μέτρων, την ε, αναγκαιότητα χρηματοδότηση ορισμένων πολιτικών και μέσω τη προσθέμενη αξία και τη στρατηγική για το 2020 θέλω να δείξω ότι υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε και να ζητήσω ε, από μια συνάδελφο από το προσωπικό. Ε, κάτι που μου είπε μάλλον, ε, τελικά χρειαζόμαστε μια πλούστευση, ναι, γιατί δεν είναι αποτελεσματική σε κοινωνικές δαπάνες. Ξέρετε, εμείς περιμέναμε μια πρόταση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απλούστευση τη διοικητική εδώ και μήνες. Είμαστε στο Μάρτιο, ακόμη δεν έχει έρθει αυτή η πρόταση. Κάποια στιγμή ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο προς τις τροπολογίες μέχρι τώρα. Ε, εδώ κάνουμε μια πολιτική δήλωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη απλούστευση. Όμω δυστυχώ δεν έχουμε ακόμη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Σαλοδόρ. Σαλοδόρ, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχει άγχο. Στην Ευρώπη είμαστε. Στι Ηνωμένε Πολιτείε μόνο πυροβολούν τον πιανίστα. Μόνο οι Αμερικανοί. Εδώ ισχύει αυτό που λέμε στη Γερμανία. Δώσε στον πιανίστα κι άλλη μια μπύρα. Αυτό είναι όλο. Ξέρω ότι λένε οι συνάδελφοι, ναι, είναι μάλλον συντηρητική η έκθεση, είναι ο ελάχιστο κοινό παρονομαστή και το καθεξή. θα έπρεπε, θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο να βρούμε τον μέγιστο δυνατό διαιρέτη. Αυτό είναι εύκολο να τον βρούμε, κανένα πρόβλημα. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, με το ελάχιστο κοινό παρονομαστή πάλι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση, μια εξαίρετη βάση για την περαιτέρω δουλειά μα, ανεξαρτήτω του τι ενδεχομένω ακούστηκε σε κάποιε παρεμβάσει. Αυτά. Για να περάσουμε λοιπόν τώρα στην δεύτερη φάση, όπου έχουμε ορίσει πως θα ασχοληθούμε πρώτα με το, η γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση, ε, διαβίου μάθηση, κοινωνικές πολιτικές. Δεύτερο τμήμα λοιπόν το οποίο για να ξέρετε τι θέματα έχουμε. Το δεύτερο τμήμα αυτού της δεύτερης φάσης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, γεωργία, αλληλεία, ε, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, μεταφορές. Αυτές είναι τα ψηλά που λέμε έτσι. Μετά έχουμε τη συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση, οικονομική Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τέταρτο τμήμα, ηθαγένεια, ε, χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, Ευρώπη στον κόσμο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Πολιτική Γειτονίας και Ανάπτυξης. Και τώρα θα έλεγα να μην περάσουμε πάλι σε γύρω συστήσεως με τους τουριστές από τις ομάδες πρώτα κτλ. Απλώς ο καθένας στον τομέα που τον ενδιαφέρει να ζητήσει το λόγο και γι' αυτό παρακαλώ ξεκινώντας να μας επισημαίνετε, να σηκώνετε το χέρι να μας δείτε πού θέλετε, σε ποιο κομμάτι θέλετε να μιλήσετε. Η κυρία Κρέλ, τρίτο τμήμα φαντάζομαι. Γκεμπράντι, δεύτερο. Γιώργνησιν, δεύτερο τμήμα. Κύριο Σταυρακάκης, για το τρίτο φαντάζομαι, έτσι. Για το τρίτο τμήμα, κύριο Σταυρακάκη. Συνοχή επίσης, τέταρτο, μάλιστα, αρκετή βλέπω. Γκοντμάνης. Τρίτο τμήμα, τρίτο τμήμα, συνοχή. Συνοχή επίσης, μάλιστα. Κύριο Φέρμ για την εξωτερική. Ε, εντάξει, είμαστε το 3 εσείς μάλιστα. Πολύ ωραία. Ich der wird gerade bei Νομίζω ότι το ΕΛΚ ακόμη πραγματεύεται εάν πρόκειται να πει κάτι ο Ζωσέ Μανουέλ Φερνάντε και τι. Κατάλαβα καλά. Ε, ναι, θέλουμε να κλείσουμε τον κατάλογο για να ξέρουμε πόσο χρόνο θα έχουμε για το κάθε κομμάτι. Συνόχι, ωραία, εντάξει. Τι ήθελες, Φρανκ. Βιώσιμη ανάπτυξη, ωραία, στο δεύτερο. Ωραία, ας ρίξουμε λοιπόν πολύ γρήγορα μια ματιά στον κατάλογο των ομιλητών. Αυτοί είναι όλοι. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτο τμήμα. Σαλβαδόρ, θες κάτι να πεις εισαγωγικά. Με μία μόνο μιλήτρια ξεκινάει το πρώτο τμήμα. Αλλά εσύ κάνεις τους άλλους την εισαγωγή στο θέμα. Γνώση για ανάπτυξη και απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. μια πιο λεπτομερή αλλά πολύ συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης. Είμαστε στη σελίδα 9 της εκθέσεως από το 29 και μετά, 10 στο ελληνικό κείμενο, πολιτικές προτεραιότητας, όπου έχουμε στην έκθεση δύο καθαρούς τίτλους. Ο ένας είναι προϋπολογισμός που υποστηρίζει τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ο δεύτερο τίτλο, ένα προπολογισμό που στηρίζει την οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι και οι δύο τίτλοι είναι θέματα που έχουν προξενήσει πολλές συζητήσεις, μερικές φορές και διαφιλονικούμενα που έχουν όμως πολύ μεγάλη σημασία ποιοτική, ιδιαίτερα εν ώψη και των ε, τωρινών δημοσιονομικών πολιτικών που δεν είχαν λάβει υπόψη την στρατηγική του 2020 γιατί δεν υπήρχε και επίσης γιατί δεν μπορούσαν να έχουν προβλέψει και την οικονομική κρίση που μας ταλανίζει και που μέσα σε πολύ λίγους μήνες μας έφεραν σε επίπεδο να συζητούμε για οικονομική διακυβέρνηση και μέτρα οικονομικού συντονισμού που εδώ και λίγο καιρό δεν θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ούτε πολιτικά ούτε σε άλλο επίπεδο. Πέραν ίσως των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαρκώς αγωνίζονταν για αυτόν τον οικονομικό συντονισμό. Ε, γνώση λοιπόν για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μας απασχολεί, το συζητούμε από το άρθρο ή την παράγραφο 37 της εκθέσεως με τη δομή που προτείνουμε ευθυγραμμισμένη στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 όπως την έχουν συζητήσει και εγκρίνει τα τρία θεσμικά όργανα. Για να ξεκινήσω, να σας πω ότι η στρατηγική για την Ευρώπη το 2020 βασίζεται σε ορισμένες θεματικές πρωτοβουλίες που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί από τη σκοπιά του προπολογισμού και αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, μιλάμε για μία δομή για την οποία πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ούτε καν τους στόχους χρηματοδότησης που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι δύσκολο για μας, αλλά Αυτές τις θεματικές πρωτοβουλίες ε, τις έχουμε θεωρήσει ως θεμελιώδες ε, προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που θα χρηματοδοτηθούν στους τομείς και στους υποτομείς για την έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε καταρχήν την αναγκαιότητα να πετύχουμε ένα 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω της Ένωσης για την Καινοτομία είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να τεθεί ε, να γίνει μια προσπάθεια γι' αυτό γιατί πολλά κράτη δεν έχουν φτάσει καν στο 2% του έκτους για την έρευνα και την εντομία και να περάσουν από το 2% στο 3% μάλλον ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει πολύ σημαντική συγκέντρωση πόρων και αυτό θα έχει πολιτικές συνέπειες. Έτσι λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο και είναι η πρώτη φορά που ζητάμε εδώ μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, χρηματοδότηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, κυρίω μέσω του 8ου προγράμματος ε, πλαισίου. Ξέρετε ότι ε, στο 7ο είχαμε 50 νης και ήταν επιτυχές και για να πετύχουμε το στόχο του 3% πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του 8ου προγράμματος πλαισίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσω μιας πιο προσανατολισμένης διαδικασίας προς τα αποτελέσματα, μέσω της απλούστευσης των ε, καινοτόμων ε, χρηματοδοτικών διαδικασιών. Όμως χρειάζεται μια πολιτική δήλωση για να αυξηθεί το ε, κονδύλι για το θέμα αυτό το ίδιο και για την καινοτομία ε, δηλαδή να δούμε για το πώς θα τεθούν σε εμπορία τα αποτελέσματα, τα επιτεύγματα της έρευνας και της καινοτομίας, ε, οπισθοδρομή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε καλοί στην έρευνα, είμαστε πολύ καλοί στην ανάπτυξη, αλλά πιθανότατα έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε στην καινοτομία. Και έτσι είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλους τομείς ε, της παγκόσμιας οικονομίας και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το τονίσει αυτό, να δώσει έμφαση. Συνεχίζουμε να ζητάμε να βελτιωθεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας ε, και ε, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας θα πρέπει να διευρυνθούν θεαματικά για την επόμενη περίοδο Πιστεύω ότι η γνώση για την ανάπτυξη και για την γενοτομία θα γίνει μέσω της ενδυνάμωσης της βιομηχανίας και των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο, στην καρδιά της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Επίσης υπάρχει μια θεματική πρωτοβουλία που είναι ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την παγκοσμιοποίηση και εκεί δεν έχουμε ποσοτικοποίηση στον προπολογισμό όμως ε, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον και το ίδιο ισχύει και για την επέκταση του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομία ε, και του μηχανισμού χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων για να προωθηθεί η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην καρδιά, όπως σας είπα, της στρατηγικής για το 2020. Αναφέρω το ψηφιακό θεματολόγιο, και προσδίδω σε αυτό ιδιαίτερη σημασία. Εδώ πρέπει να γίνουν επενδύσεις ε, για την υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου, κυρίως ε, όλα όσα αφορούν ε, την επέκταση το εις Έχουμε πει ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη την οικονομική, την ανάκαμψη της οικονομίας και θέλουμε να φτάσουμε το όσο περισσότεροι πολίτες, κυρίως στις λιγότερα αναπτυγμένες περιοχές, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Επίσης, εδώ πρέπει να τεθούν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ουρανό και το διάστημα. Τόσο τα συστήματα πλοήγησης όπως το Γαλιλαίο, όπως ε, και το σύστημα του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού που θα δημιουργήσουν πολύ σημαντικές οικονομίες κλίμακας χρειάζονται επενδύσεις. Ξέρετε ότι έχουμε χρηματοδοτήσει τα διαστημικά προγράμματα ε, δορυφορικής πλοήγησης μέσω του συστήματος ευελιξίας που δεν μας ε, χρησιμεύει για το μέλλον, δηλαδή ε, κάναμε όλες αυτές τις επενδύσεις, ε, αλλά όχι με τον πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την παράγραφο αυτό που λέγεται ότι χρειάζεται ε, ε, εργατικό δυναμικό που θα έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Σε αυτά τα αναφέρω στις παραγράφους 45 και 46, γιατί στην ίδια τη στρατηγική για το 2020 υπάρχουν ε, αυτά τα benchmarkings και πρέπει επίσης να αφιερώσουμε τα περίπτωτα κονδύλια και σε αυτούς τους τομείς. Εδώ θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αναφέρεται στο 46. Δεν έχουμε βέβαια έναν εξαντλητικό κατάλογο. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα αναφερθούν στο θέμα αυτό και μέσω τροπολογιών αλλά τέλο πάντων ε, για να μην είναι ατέλειωτη η εκθεσή μου έπρεπε να επικεντρωθώ σε ορισμένε προτεραιότητε. Σα ευχαριστώ και πριν περάσουμε τώρα στου ομιλητέ για το πρώτο τμήμα, για το πρώτο μέρο, για την γνώση δηλαδή, για την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα ήθελα να ζητήσω από δύο ομάδε, μάλλον τρει ομάδε, οι οποίε δεν έχουν ζητήσει το λόγο. Το Ρίτσαρτ να ζητήσω, να ρωτήσω, θέλει να μιλήσει για κάποιο θέμα, όχι. Οι πράσινοι θέλουν το λόγο για κάποιο από τα ζητήματα. Ιζαμπέλ. Ναι, μα βάλτε ακουστικά. Βάλτε ακουστικά σου, Ιζαμπέλ. Δεν έχω κανέναν ομιλητή για κανένα από τα τμήματα, ούτε για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο από τους πράσινους. Θα ήθελαν οι πράσινοι να πάρουν το λόγο για κάποια από αυτά τα τμήματα αυτά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι υποχρεωτικό άλλωστε. Μιγγέλ. Για αυτό το θέμα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άρα θα συνεχίσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο επόμενος ομιλητής τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Σαλβαδόρ. Γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά εξαντλητικός ο κατάλογος των θεμάτων που αναφέρονται. Όταν καταρτήσαμε την έκθεση και όταν αρχίσαμε τις... Ε, όταν θα αρχίσουμε τελικά τις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να δούμε ποιες, ποιοι τομεί είναι πραγματικά πραγματικής προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι σε θέματα ερευνά, σε θέματα καινοτομία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατρανώσει τη φωνή του, γιατί θα δυσκολευτούμε να βρούμε μεμονωμένε χώρες που θα πολεμήσουν με τα θέματα αυτά. Ο Σαλβαδόρα ανέφερε ότι θα πρέπει να βάλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προσπαθειών. Συμφωνώ. Αλλά επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλουμε και την αριστεία στο επίκεντρο της πολιτικής. Αριστεία σε επίπεδα έρευνας και εντομίας. Δύο τομεί θα ήθελα να υποδείξω. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο είναι ακόμα περιορισμένο σχετικό. Και νομίζω όμως ότι η ανεξάρτητη έρευνα είναι πολύ σημαντική. Είχαμε και τον πρώτο βραβευμένο με βραβείο Νόμπελ από το πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να το ενισχύουμε. Αυτό εννοώ αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο τομέα το, του IT, που ήταν ιδέα και του κυρίου Μπαρόσο. Πολλοί στο Κοινοβούλιο ήμασταν κάπως σκεπτικοί, γιατί θεωρούσαμε ότι αφαιρούσαμε απλά χρήματα από την καινοτομία χωρίς ε, να υπάρχουν νέα κονδύλια. Αλλά νομίζω ότι σε πολλούς κλάδους μπορούμε να βάλουμε μαζί την έρευνα και την καινοτομία για να βρούμε νέα κονδύλια για το IT, για την ε, τεχνολογία πληροφορίας. Και αυτό σαφώς και θα υπογραμμίσει πιο πολύ την καινοτομία και τα προγράμματα πλαίσιο μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Είδαμε ότι 70% ήταν η αύξηση κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, άρα αυξήθηκε σημαντικά. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ισχυροί στον τομέα αυτό. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική για το διάστημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο, θα πρέπει ασφαλώς να συνεχίσουμε να βρίσκουμε κονδύλια και από άλλα προγράμματα. Να έχουμε σίγουρα αρκετά κονδύλια για τα προγράμματα αυτά, τα οποία πραγματικά είναι ευρωπαϊκά στη φύση τους. Ευχαριστώ. Ράιμα Μπέγκε τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο εισηγητής κατέρτισε ένα καλό κείμενο στο κεφάλαιο αυτό. Συμφωνώ με την Αν ότι ήταν μεγάλη ε, ο σκεπτικισμός ε, για το κατά πόσο θα υπήρχε ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την τεχνολογία της πληροφορίας με το IT. Αυτό φαίνεται ότι πάει μια χαρά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο έντονα και να αναφέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να κληθούν μαζί με τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν ένα δικό χάρτη για το πώς και πότε θα καταλήξουμε στο 3%. για την ε, προώθηση των ε, ε, επενδύσεων των ιδιωτικών, για το πού μπορούν να υπάρξουν συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και τομέα και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση. Να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή και να δούμε και τι θα γίνει και με την Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο και με τους εθνικούς προπολογισμού. Σύμφωνο για την έρευνα και την καινοτομία υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη, αλλά έχουμε το πρόβλημα ότι η έρευνα δεν κινείται στον πράσινο τομέα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτό που έκανε και ο Σαλβαδόρ και η κυρία Καρβάλιο παρουσίασε σε ό,τι αφορά την απλοποίηση των ε, ε, διαδικασιών και εδώ απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να γίνει για την κατεύθυνση αυτή πρωτού να, να πανίσουμε πιο πολλά κονδύλια. Και θεωρώ ότι είναι σαφές ότι τα προγράμματα διαβίου ε, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή διάσταση της απασχόλησης. Ε, το πώς χωρίς να ενσωματωθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο θέμα της ευρωπαϊκής έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το αναφέρει ο Σάλβαδορ. Το τι κάνουμε με τα μεγάλα project, τα οποία κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα και πάντα χρειάζονται επιπλέον πόροι τελικά στο τέλος του χρόνου. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πέρα από το 2020 είτε θα το κάνουμε αυτό ή θα βγουν αυτά τα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή ή θα ψηφιστούν αυτή, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό των προγραμμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Γιώραν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο που θα μιλήσει για την ομάδα μα δεν ε, έχει καταφέρει να έρθει, οπότε θα μιλήσω εγώ εκ μέρου του. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα. Και θυμάμαι πολύ καλά το δημόσιο διάλογο που είχε αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάνα δύο χρόνια με ε, στόχο τον προσδιορισμό των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών και ήταν ξεκάθαρο πως όλοι, εθνικά κοινοβούλια, ε, εκπρόσωποι των κλάδων κτλ, εμπλεκόμενοι φορείς, συμφωνούσαν ότι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητα είναι ακριβώς αυτή η έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη. Βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα την ορίσουμε και βέβαια πώς θα εστιαστούμε στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, εκεί που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνο στα κράτη-μέλη. Πρέπει δηλαδή οι πόροι μας να συντονιστούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Επίσης θα πρέπει να βρούμε και τα κατάλληλα μέσα, γιατί βέβαια η υπεροχή είναι καλό στόχος, αλλά δεν μπορούμε μόνο να στηριχθούμε στην Οξφόρδη και το Κέμπριτζ ή τη Λόβερ και το Παρίσι. Πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό στα ανατολικά κράτη της Ευρώπης ή στα φτωχότερα κράτη. Πρέπει και εκεί να βοηθήσουμε και να αναπτύξουμε τρόπους αξιοποίησης πολιτικής συνοχής για την καινοτομία, για την προηγμένη εκπαίδευση. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τις πιο αδύναμες περιοχές μόνο με Το άλλο, το, άλλωστε το υποστήριξε ο κύριο Μπαρόσο, το έλεγε πριν από κάνα δύο χρόνια. Υπάρχουν εκατοντάδε χιλιάδων Ευρωπαίων ερευνητών που φεύγουν στις ΗΠΑ γιατί βρίσκουν καλύτερε επιλογέ. Και όχι μόνο επιλογές yes, έρευνας, αλλά και επιλογέ ή εναλλακτικέ καινοτομία και επιχειρηματικές. Και, γι αυτό, και εκεί πάλι πρέπει να δώσουμε έμφαση για να ξανακρατήσουμε την έρευνά μα μέσα στην Ευρώπη για του ερευνητέ. Ακόμη κάτι άλλο, Σαλβαδόρ είπε ότι έχει ένα εξαιρετικό κατάλογο διαφόρων θεμάτων. Αλλά νομίζω ότι έχει ξεχάσει κάτι από τον εξαιρετικό. Το πιο, τα πιο κοινωνικά προγραμμα, ε, προσανατολισμένα προγράμματα, πρόοδο για την πρόοδο και ούτω καθεξής, δεν τα κάνουμε για το μέλλον. Πρέπει να είμαστε σε θέση να μη λησμονήσουμε την πολιτική ή τη διάσταση, την συνεκτική της ενσωμάτωσης αυτών των πολιτικών που μπορούν να διαδραματίσουν αυτές τις πολιτικές για την Ευρώπη και επίσης χωρίς να έχουμε καταλήξει σε μια οριστική θέση, έχουμε συζητήσει το θέμα της έρευνα στην ε, πολιτική μου ομάδα έτσι και καταλήγουμε ότι θα πρέπει τα προγράμματα όπως Ήτρα και Γαλιλαίος να τα χειριστούμε έτσι, να αναπτύξουμε μια μέθοδο ώστε αυτά να μην αποβαίνουν πάντα ει βάρο των άλλων προγραμμάτων. Να μην τρώνε δηλαδή κονδύλια πάντα από τα άλλα προγράμματα. Είναι προγράμματα μακροπρόθεσμα, μεγάλα προγράμματα υποδομών και όπω είπα δεν έχει κλείσει η συζήτηση στην πολιτική μου ομάδα και απλώ θέτω το θέμα προ συζήτηση εδώ. Πρέπει να βρούμε δομέ, ενδεχομένω με χωριστέ ε, θέσει στον προπολογισμό, ώστε να μην τρώνε τα κονδύλια από τι άλλε ε, ε, πολιτικέ. κύριος Πόρτας. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το τομεί μπορούμε να έχουμε σημαντική σύγκληση. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν του προηγούμενου ομιλητέ. Το πρόβλημά μου, η άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξή. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ποιοτικά ζητήματα, γιατί εγώ νομίζω ότι εδώ μπορεί να αποκλίνουν οι απόψεις μας. Νομίζω ότι η τάση της έκθεσης είναι ουσιαστικά κάπως ε, προς την κατεύθυνση ότι για την έρευνα και την ανάπτυξη το ουσιαστικό είναι η ανταγωνιστικότητα και η αριστεία. Δηλαδή έχουμε δύο μαχικές λέξεις εδώ που όμως έχουν και μια συνέπεια. Μόλις εργαστήκαμε στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης ε, ακριβώς για να έχουμε την διάσταση της εφαρμογής. Και αυτό είναι το πρώτο. Σίγουρα χρειαζόμαστε εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση εξ ονόματος, ε, μάλλον ονόματι της ανταγωνιστικότητας να περιορίσουμε την ζωτική έρευνα, τη θεμελιώδη έρευνα και τελικά να έχουμε μια έρευνα που δεν θα είναι ούτε θεμελιώδης ούτε εφαρμοσμένη. Δηλαδή πρέπει να δούμε ε, πώς ε, διαφοροποιούνται αυτές οι δύο κλασικές μορφές έρευνας. Η πρότασή μου για το κείμενο θα είναι να εργαστούμε επί αυτού του θέματος και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε καλά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης ανάλογα με τα διάφορα είδη έρευνας. Γιατί μπορεί η έρευνα να υποστηρίζεται βασικά από την αγορά, υπάρχει όμως και άλλη είδους έρευνα που ε, είναι πιο ε, επικίνδυνη και υπάρχει και άλλη, δηλαδή θέτει περισσότερους κινδύνους και υπάρχει και άλλη έρευνα που είναι δημόσιας χρηματοδότησης, δημόσιας φύσης. Έχουμε και ένα πρόβλημα κρυφής ε, υποχρηματοδότησης σε κάθε ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα και πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνθήκε εργασία των νερών ερευνητών. Όταν ε, μιλάμε για την αναγκαιότητα να αυξήσουμε τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη, πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουμε ένα θέμα κρυφής υποχρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μα, γιατί ε, πρέπει ο ερευνητής να ε, βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση οικονομικά για να κάνει και ποιοτική έρευνα. Το επόμενο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι το εξής. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων η επιστημονική έρευνα εξαρτάται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε άλλες χώρες ε, υπάρχουν πολλά μεγάλα προβλήματα για την έρευνα. Θα ήθελα και μία αναφορά σε αυτή την πτυχή, γιατί νομίζω ότι αυτό προσανατολίζει τις εργασίες. Και για τα μεγάλα προγράμματα, για το Γαλιλαίο, τι να σας πω, έχω κάποιες αμφιβολίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε διεθνείς λύσεις συνεργασίας για αυτά τα μεγάλα προγράμματα, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να κάνουμε και εξοικονόμηση. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Τζοχά. Νομίζω ότι α, μπορώ να συμφωνήσω με το είπαν ο κύριο Φέρμ και ο κύριο Πόρτα τώρα. θα ήθελα εκ μέρου τη ομάδα μου να υπογραμμίσω κάτι το πολύ, ουσιώδους, το πολύ ουσιώδες. Μετά όσα συμβαίνουν και εξακολουθούν να συμβαίνουν τώρα στην Ιαπωνία, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να συζητούμε εν γέννη τα θέματα τη ανανεώσιμη ενέργεια. Πρέπει να καταστεί προτεραιότητα υπαριθμών 1 και όλα τα ζητήματα τη αποτελεσματικότητα τη χρήση τη ενέργεια και των, απο... Ε, ανανεώσιμων μορφών πρέπει μέσα στην έκθεση και στι συστάσει μα να προσλάβουν μία ε, πρωταρχική θέση Έστω και χρειαστεί να συζητήσουμε υπό του όρου του κύριου Έτσιγκερ, που είπε ότι είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε τι θέσει μα περί πυρηνικών. Και ενδεχομένω και να συζητήσουμε το πρόγραμμα ITER και το πόσο κοστίζει στον προπολογισμό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αποτελεσματικότητα πρέπει να έχουν κύριο ρόλο στην έρευνα. Και για το Γαλιλαίο. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό φυσικά. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να, να μετριάσουμε τον προπολογισμό του, να μην ε, απορροφά όλα τα κορδίλια. Γιατί είπαμε το smart μερικές φορές είναι και small, δεν είναι απαραίτητα big. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τάση συνήθως να χρηματοδοτούμε τα μεγάλα ε, σχέδια, τα μεγάλα έργα και να λησμονούμε ότι και τα μικρά μπορεί να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και εν πάση περιπτώσει να μην λησμονούμε ότι χρειάζεται πάντοτε να δίνουμε την έμφαση στην αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας. Ε, έστω και στα παλιότερα προγράμματα δηλαδή ή έργα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες προσπάθειε να μένουν οι ερευνητές και για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη, να μένουν εδώ και σε τελευταία γιατί να μην, πηγαίνουν, ε, να μην πηγαίνουν από τη μια στην Οξφόρδη και από την άλλη μόνο στη Φίσερ, να υπάρχουν και, άλλοι, και άλλε λύσει. Όπως είπα, πρέπει να εμπνευστούμε από αυτά τα γεγονότα που δυστυχώς δραματίζονται σε ζωντανό χρόνο ε, και να μην παραμένουμε στο business as usual. Ευχαριστώ. Κυρία Καμπάγια τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω, όπως και οι συνάδελφοι, τη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης της καινοτομία στην Ευρώπη, ολόκληρη και υπογραμμίζω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είπαμε ότι το FTF είναι ένα πολύ σημαντικό ταμείο, ε, ένα πολύ σημαντικό μέσον και χαιρετίζω την ε, σημείωση στην ε, έκθεση του κυρίου Γαρίγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο να το υποστηρίξουμε περισσότερο. Ναι, λοιπόν, στηρίζει την καινοτομία, αλλά μου ότι θέλουμε αυτό το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο να αποτελέσει και την βασιλική οδό για την υπεροχή, να χτίσει δηλαδή τους όρους και τα θεμέλια για την οικοδόμηση της ε, έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπα, βασιλική οδός και θεμέλια. Και επίσης δεν μπορούμε στα διαρθρωτικά ταμεία να επιτρέψουμε να λησμονούνται στο κοινωνικό, το κοινωνικό ή τα διαρθρωτικά δεν μπορούν να λησμονούν τις υποτροφίες, την δυνατότητα οι επιστήμονες, οι φοιτητέ, οι μηχανικοί που ενδεχομένω χρειάζονται περισσότερο έρευνα να αξιοποιούν αυτά τα ταμεία. Και επίσης, όπως είπα, χρηματοδότηση δεν μπορούμε να έχουμε κατάλληλη εάν δεν υπάρχουν απλοί κανόνες, απλούστευση. Η απλούστευση, όπως λέμε πάντα, είναι η πιο σημαντική πτυχή που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε. Ιδάλλως δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε σωστά τη χρηματοδότησή μας. Χρειαζόμαστε πιο απλούς, πιο αποτελεσματικούς κανόνες και στην έρευνα και στις υποδομές. Έτσι ώστε να μπορούμε κατά τρόπο απλό, αποτελεσματικό, διαφανή να εκτελούμε τα έργα για την έρευνα και την κοινοτομία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ζαρβαδόρ, θε να πει κάτι για να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι ή θέλει να αρχίσει αμέσω την εισαγωγή σου του δεύτερου, για το τρίτο κομμάτι. Όχι, για να κλείσουμε αυτό το σημείο. Πριν να, να ξεκινήσω το επόμενο, να υπενθυμίσω στη συνάδελφο ότι για το θέμα της ενέργειας θα μιλήσουμε στη συνέχεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να πω ότι διαπιστώνω τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων που πήραν το λόγο σχετικά με την αναγκαιότητα να θέσουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και την έρευνα στο επίκεντρο της γνώσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν ένα από τα καλύτερα ε, πράγματα τα οποία έγιναν κοινωτικές δαπάνες ε, και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Προσταμένης Αξίας ε, με την εφαρμογή στις πολιτικές μας δίνουν ένα καλό εργαλείο ανάλυσης. Εγώ, παραδείγματο χάρη, είδα την εκτέλεση ε, και είδα πώς ακριβώς ε, στην ε, Ισπανία δαπανήθηκαν τα χρήματα από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και πραγματικά με εξέπληξαν τα αποτελέσματα. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλή πολιτική έρευνα σε κοινοτικό επίπεδο και φυσικά δεν υλοποιείται μόνο μέσω του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου, αλλά και μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και των νέων μέσων ε, που αποκτήσαμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Υπάρχει όντως ε, αυτή η καλή ερευνητική πολιτική και τελικά προκύπτουν και τα αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αντιογωνιστικότητα. Εγώ επιμένω. Τώρα, και αυτό πρέπει να το αντικατοπτρίζουμε ε, στην έκθεση. Τι μας διαφοροποιεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα αν είναι καλύτεροι ερευνητέ μας ή χειρότεροι. Ε, εγώ νομίζω ότι η ευρωπαϊκή έρευνα βρίσκεται σε πρώτο επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα της καινοτομίας ως ε, ένα διεύλο να φέρουμε στην αγορά όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα των ιδρυμάτων μας. Τελικά, στην ε, βάση όλη τη έρευνα υπάρχει ένας νεαρός ερευνητή και θέλουμε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορεί να ε, επιβιώνει αξιοπρεπώς. Αν ε, αυτός ο νέος ερευνητής δεν βρίσκεται μόνο σε μια ιδιωτική εταιρεία στη Siemens, χάρη, αλλά και σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Ε, στα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη. Και χωρί αυτό το νεαρό ερευνητή δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική ερευνητική πολιτική. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πλοκό το ζήτημα. Άκουσα τι είπε και η συνάδελφο Καρβάγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αριστεία, αλλά και ο οδό προ την αριστεία. Η αριστεία δεν είναι μόνο ένα θέμα που θα πρέπει να επικεντρωθεί η έρευνα, δηλαδή να επικεντρωθούμε συγκεκριμένου τομεί που είναι πολύ ανταγωνιστική, πρέπει να γίνεται η έρευνα σε όλους ε, ε τους τομείς ε, και μάλιστα πρέπει και τα διευθυντικά ταμεία να προσανατολίζονται προς αυτή την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφή οδικό χάρτη, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πώς θα φτάσουμε στο 3%. Αυτό το 3% στην έρευνα ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση, αλλά και στην προσπάθεια που θα καταβληθεί, όχι μόνο από τις χώρες, αλλά και από την κοινότητα. Δεν μπορούμε να μόνο με ένα απλό benchmarking να προσπαθήσουμε από το 2 να φτάσουμε στο 3%. Αυτό το 1% αύξηση προϋποθέτει πολύ σημαντική αλλαγή στις πολιτικές και πρέπει να έχουμε προκαταρτήσει, προκαταρτήσει πολιτικές, να έχουμε εκταμιεύσει πόρους ε, για ερευνητικά ζητήματα. Εμείς ε, με αυτό ξεκινάμε, λέμε ότι συμφωνούμε με το 3% γιατί αυτές οι αποφάσεις είναι θεσμοί που πρέπει να τις πάρουν. Όμως ε, μπορώ να σας πω ότι αυτό το 3% έχει άμεση επίπτωση στους προϋπολογισμούς της Ένωσης και θα πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Σας είμαστε εδώ ρεαλιστές, σας γνωρίζουμε όλοι τι υπάρχει πίσω από αυτό και τι προσπάθειες επενδυτικές θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον για αυτό το 3%. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση στο σημείο αυτό και είμαι... Σίγουρο ότι με τι τροπολογίε που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι θα εμπλουτιστεί το κείμενο. Σαλβαδόρ, να πάρεις μια ανάσα και μετά να κάνεις μια εισαγωγή κατευθείαν αν θέλεις στο δεύτερο τμήμα, τη δεύτερη φάση. Για την βιώσιμη ανάπτυξη, ε, γεωργία, αλληλεία, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, πολιτικές για τις μεταφορές. Έχουμε κατάλογο ομιλητών. Τσέσλαβ Σικιάσκι Φρανκ Έγγελ και Μπρίτα Ραϊμας, Ισαμπέλ Ευχαριστώ. Είναι ε, κάπως πιο ευρύ το θέμα αυτό, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές διαφορετικές πολιτικές και τίτλους. Ε, βέβαια έχουμε και ορισμένες ε, αντιφάσεις εδώ. Τώρα, η βιώσιμη ανάπτυξη. Στην σελίδα 11 του αγγλικού κειμένου σελίδα 13 του ελληνικού, Έχουμε εδώ την κάλυψη της κοινή γεωργικής πολιτικής από τις παραγράφους 47 μέχρι 51. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να συνεισφέρει ε, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη για το 2020, αν και φυσικά έχει και ξεχωριστούς στόχους από αυτή τη στρατηγική. Για μας η κοινή γεωργική πολιτική βρίσκεται παγιωμένη στη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας είναι αυτή που προσδιορίζει τους στόχους της και τα καθήκοντά της. <clears throat> Υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα τον πολυλειτουργικό ρόλο της ε, ΚΑΠ ως μια πολιτική που θα παρέχει δημόσια αγαθά πέρα και των γεωργικών αγορών. Και αναφέρομαι κυρίως ε, στο θέμα της επισητιστικής ασφάλειας, την διατήρηση της υπαίθρου, την ε, ποικιλομορφία, τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της επικρατείας μας, βελτίωση της βιοποικιλότητας και της ε, ευημερίας των ζώων. Της καλής διαβίωσης των ζώων και φυσικά έχει αντίκτυπο, μπορεί να έχει αντίκτυπο κοινή γεωργική πολιτική και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί οι πολλαπλοί στόχοι που περιλαμβάνονται στην ε, αναθεώρηση της ε, ΚΑΠ, από την ε, οποία, για την οποία ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει και συγκεκριμένες προτάσεις επόμενους μήνες, μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι δεν βλέπουμε δυνατό να μειώσουμε τον προϋπολογισμό για την ΚΑΠ την επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Αλλά το αντίθετο, αν θέλουμε μια βιώσιμη τέτοια πολιτική που να μπορέσει να πληρώσει τους στόχους της, που έθεσε και ο Επίτροπος, θα έπρεπε να έχουμε πιστώσεις παρόμοιες με αυτούς που είχαμε για το 2013. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε για επίπεδο χρηματοδότησης παρόμοια με αυτή που έχει η κοινή γεωργική πολιτική για το 2013. Θα μπορούσαμε να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις ε, και τις άμεσες πληρωμές στο δεύτερο πυλώνα. Επίσης ε, πιστεύουμε ότι το διαρθρωτικό ταμείο ε, που έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να είναι ιδιαίτερα συντονισμένο στη λειτουργία του με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και φυσικά στη δομή του πρέπει να περιλαμβάνει την διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αλία τώρα. Έχουμε μια κοινή ελευτική πολιτική η οποία λειτουργεί σχετικά καλά. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι στις ε, παράκτιες περιοχές χρειάζεται μία ε, ισχυρή ελευτική πολιτική για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Είναι δύσκολο να βρούμε εναλλακτικέ. Έτσι λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε μια κοινή ελευτική πολιτική που να είναι αηφόρος, να διατηρηθούν ε, ή τα αποθέματα των ηχθείων, αλλά να υπάρχει και μια δομή έτσι ώστε ο λευτικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικός και πηγή απασχόλησης και πλούτου. Τώρα, το θέμα της κλιματικής αλλαγής ε, και της επάρκειας των φυσικών πόρων. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα επίμαχο σημείο. Από τη δική μου σκοπιά, πέρα από το ότι ήδη υπάρχουν ε, γραμμές του κοινωτικού προπολογισμού που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, Εμένα οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, ο όρος κλειδί είναι το mainstreaming, δηλαδή η συμπερίληψη σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ένωσης. Οι δράσει για το κλίμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα σχετικά κεφάλαια των κοινοτικών δαπανών. Εδώ επιζητούμε την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Είναι ένας από τους κύριους στόχους τα κριτήρια της ε, εφορίας, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και της ενεργικής αποδοτικότητας βρίσκονται στη στρατηγική για το 2020. Αν υιοθετήσουμε αυτή τη στρατηγική, υιοθετούμε και τους ενεργειακούς στόχους. Επίσης υπάρχει και εδώ ένα φλάξι, μια θεματική πρωτοβουλία ε, για τους αποτελεσματικούς ε, πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ενεργειακά. Δεν έχουμε ούτε εδώ ποσοτικοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, αν σε κάτι όλοι συμφωνούμε, είναι ότι ε, το τμήμα της ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, δηλαδή πρέπει να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση, πρέπει να έχουμε αύξηση εδώ. Αυτό είναι κλειδί για την ε, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και είναι και κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ευρώπη το 2020. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο πολιτικού συντονισμού και η χρηματοδότηση της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να γίνει μέσω του σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών, του σχεδίου ΣΕΤ. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη, αυτό θα το διασφαλίσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα Ξέρετε, αυτό είναι από το σημείο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πιο επικλητικό στις τρέχουσες δημοσιονομικές προεπτικές. Είχαμε μία ποσότητα στο πακέτο πρώτη που μειώθηκε ε, περισσότερο από το ίμιση και αυτό είχε πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις όταν ε, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα επικοινωνιών και κυρίως ε, όταν μιλάμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Δεν είχαμε επαρκές επενδύσεις, ενώ τώρα πρέπει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις σε δίκτυα, να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Εδώ αναφέρονται κάποια αριθμητικά στοιχεία, αδύνατα να μεταφραστούν. Τρίλιον euros λέει ο μιλητή στα αγγλικά. Χρειαζόμαστε 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ε, βρίσκεται ούτε σε εθνικού ούτε σε κοινοτικό προπολογισμό. αυτό το νούμερο. Καταλαβαίνετε βέβαια πόσο μεγάλη πρόκληση αποτελεί για καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να συνεισφέρει εδώ ο κοινωνικό προπολογισμό. Και αυτή είναι άλλη πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Δηλαδή θα πρέπει να μεταφερθούν πόροι από άλλου τομεί ή να επαναπροσδιορίσουμε κοινωτικέ πολιτικέ έτσι ώστε το θέμα τη ενεργειακή αποδοτικότητα και των νέων δικτύων υποδομή και μεταφορών να καλύπτονται. Κατόπιν θα περάσουμε στην πολιτική συνοχή πρόεδρε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι για το σημείο αυτό ανέφερα τα κυρίε ιδέε τη έκθεση και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν και πολλέ πολιτικέ αποφάσει σχετικά. Ευχαριστώ. Κύριε Σκαμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία λεπτά. Ik zal, ik zal tempo maken. Uh, ik, ik dank Salvador Garriga. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ τον Salvador Garriga, όχι μόνο ως ε, μέλος άλλης ομάδας, αλλά και ως μέλος της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, γιατί πολλά συμπεριέλαβε από τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής μας και τις κόκκινες γραμμές ε, της έκθεσης μου, ότι πρέπει να έχουμε μόνο, όχι μόνο ηθικό καθήκον να ακολουθήσουμε την οικονομία, αλλά και πραγματικά επιτακτική ανάγκη να δούμε τι γίνεται στην Κίνα, όπου ε, υπάρχει ανταγωνισμό και στη βιώσιμη τεχνολογία. Αν δεν επιταχύνουμε λοιπόν στην Ευρώπη, δεν θα χάσουμε μόνο στους μισθούς, αλλά θα χάσουμε και ε, στην τεχνολογία γιατί σε πολλά πράγματα μας έχει ήδη ξεπεράσει η Κίνα. Να ευχαριστήσω και στην ε, έμφαση που δίνεται στα κριτήρια βιωσιμότητας σε άλλους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό το mainstreaming. Αυτό που λείπει είναι η επικέντρωση στις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις μάλιστα που έχουν αρνητικό αντικτύπο σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους βιωσιμότητας για το κλίμα, τη βιοπικιλότητα και το καθεξής. Παραδείγματα. Ε, θεωρούμε, μάλλον ε, υποστηρίζουμε τις επιδοτήσεις ε, σε εξορίξεις άνθρακα, αλληλεία. Δίνουμε μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων στην αλληλεία. Δεν είναι βιώσιμη αυτή η δομή και μας κοστίζει δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και τα στερεί από άλλους τομείς, τους οποίους θα έπρεπε να ενισχύουμε. Νομίζω λοιπόν από την Επιτροπή αυτή θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά και έχουν γίνει συμφωνίες στα πλαίσια του G20 στη Συμφωνία ε, Βιοπικιλότητας ε, την Περσινή και είπαμε ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε περιορίσει τέτοιο ποσοστό, το χύψη ποσοστό ε, βιοκαυσίμων. Ε, ορυκτών καυσίμων. Ας ε, αποτελέσει αυτό και δικό μας στόχο για την γεωργία τώρα, Πρόεδρε. Η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος απότερος στόχος για τη γεωργία είναι όχι το εισόδημα των ε, γεωργών, αλλά η ψηστική ασφάλεια. Τα χρήματα λοιπόν που έχουμε Ας τα αξιοποιήσουμε για την καινοτομία και για την βιωσιμότητα του, κλάδι, του κλάδου. Να υπάρξει και μεταρρύθμιση του κλάδου, προκειμένου μακροπρόθεσμα να πετύχουμε πολύ περισσότερο από αυτά που πετυχαίνουμε ε, σήμερα, που ουσιαστικά η πολιτική που ακολουθούμε σήμερα θέλει να διατηρήσει το status quo. Τέλος, ε, στην αλληλεία. Η παράγραφος για την αλληλεία ξεκινά με τα συμφέροντα του τομέα του κλάδου της αλληλείας στις παράκτιες περιοχές καλό και αυτό, αλλά θα ήθελα να δώσουμε έμφαση ότι αν θέλουμε η αλληλεία να καταστεί ε, αποδοτική, μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να περιορίσουμε σημαντικά την αλληλεία μας τώρα και ας χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα χρήματα που ε, δίνουμε στην αλληλεία για να αναπτύξουμε άλλες οικονομικές δραστηριότητε στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργενσεν τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τόσο υπόθηκα μόλις τώρα σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν και του στόχους και τις επιλογές δική μου έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους τομείς εκείνους όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Αυτό και βέβαια για <clears throat> λόγους διαπραγματευτικούς γιατί είναι πιο εύκολο να βρούμε επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε αυτό, αλλά και γιατί αποτελεί και μεγάλο όφελο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιβάλλον. Και οι κλιματικέ αλλαγέ βεβαίω έχουν τεράστια σημασία. Καταρχά, για ένα απλό λόγο, ότι είναι αυτά τα προβλήματα ε, φύσεως που δεν γνωρίζει σύνορα και ω εκ τούτου αν ο ένας πληγεί ο, το πρόβλημα αφορά και τον άλλον. Περιβάλλον λοιπόν και κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να εξετάζονται ως δαπάνες. Γιατί μπορεί βέβαια να έχουν ένα κόστος, αλλά τελικά όσο και να μας κοστίσουν, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας, αποτελούν τη βάση για μια υγεία οικονομία και αυτό βεβαίω το ξέρουμε εδώ και χρόνια, ταυτόχρονα όμως ε, ε, αποδεικνύει την ε, σημασία του καθώς παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση τιμές των ορυκτών καυσίμων, καθώς η σπάνιση των ε, πόρων μας ε, είναι όλο και πιο προφανής, καθώς η μεγάλη κρίση στην Ιαπωνία με τα πυρηνικά μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε το ενεργειακό μας μείγμα, καθώς η Κίνα προσδιορίζει το 12ο πενταετές της πρόγραμμα και άρα βλέπουμε κύριε Σιγητά ότι επενδύονται 3 εκατομμύρια μόνο, μόνο για τις εκπομπές. Χώρια οι ανανεώσιμες πηγές κτλ. Και αυτό κύριε εισηγητά μας δίνει διαφορετική διάσταση στο πόσο 3 εκατομμύρια θα δαπανίσουμε εμείς. Περιβάλλον λοιπόν, περιβαλλοντικές αλλαγές ή κλιματικές αλλαγές δεν είναι θέματα τα οποία, δεν είναι χρήματα τα οποία πρέπει να βγουν από άλλα κεφάλαια, να αποτελέσουν μια θυσία δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει να θυσιάσουμε κάποιο άλλο κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσουμε το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουν τη δική του χρηματοδότηση και μεγάλη χρηματοδότηση για το μέλλον. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτές, ε, αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει και χάρη στο mainstreaming, στην εισαγωγή δηλαδή των, ε, της διάστασης αυτής του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής στις άλλες πολιτικές. Βέβαια, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταχθεί αυτό μέσα στην έκθεση, αλλά δεν ξέρω πόσο λεπτομερώς. Θα το δούμε αυτό με τις τροπολογίες που πρόκειται να καταθέσουμε. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, κλείνοντας να πω ότι η μετάβαση και μια ομαλή μετάβαση ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε έννοια. Ευχαριστώ, Σικέσκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να φερθώ στην αεφορονάπτυξη, στην γεωργία έχουμε διατηρήσει δύο πυλώνες, όπου ο πρώτος καταγράφει την καλλιεργούμενη γη με το δυναμικό της, παραγωγή, της παραγωγής, της παραγωγικότητάς της και δεύτερον θα πρέπει, πιστεύω, να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες επί του περιβάλλοντος ή των κλιματικών αλλαγών της γεωργικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν Όσο πιο πράσινη, όσο πιο οικολογική γίνει η γεωργία, τόσο το καλύτερο. Χρειάζονται όμως, χρειάζεται όμως να δούμε και δύο τομείς όπου μπορούμε να ε, παρουσιάσουμε και τιμές καλές και κέρδος, κερδοφορία, δηλαδή να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητά μας, έναντι και του υπόλοιπου κόσμου. Ας δούμε λοιπόν το κόστος παραγωγής, που είναι πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη. Το 20% του εισοδήματος του Ευρωπαίου γεωργού ε, προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και είναι πολύ υψηλότερο, μάλλον είναι πολύ χαμηλότερο από το εισόδημα των λοιπόν ε, κλάδων. Ε, εξαρτάται δηλαδή από τον προπολογισμό μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβίωσή του ο Γεωργό, αλλά πάλι δεν φτάνουν αυτά. Βλέπουμε λοιπόν γιατί φεύγει ο κόσμο από τη Γεωργία, γιατί γυράσκει ο γεωργικό μα πληθυσμό και γιατί δεν έχουμε αρκετού νέου ανθρώπου μέσα στο πλαίσιο τη Γεωργία. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Η Γεωργία έχει μια πολύ σημαντική διάσταση και ένα ρόλο σημαντικό να διαδραματίσει, ιδιαίτερα στα σχετικά νεότερα μέλη κράτη-μέλη, όπου πρέπει να επιταχύνουμε τη γεωργική ανάπτυξη, να αναπτύξουμε τις υποδομές μας, την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή τα οποία σε τελευταία ανάλυση συμπίπτουν με την πολιτική της συνοχής και όπου θα πρέπει να εντοπίσουμε το τομείς στους οποίους η ανάπτυξη της υπαίθρου συνδέεται με την συνοχή και όχι κατά ανάγκη, γιατί δεν έχουμε αρκετούς ε, πόρους ε, στην κοινή γεωρική πολιτική. Αλλά μην ξεχνάμε και ποιες είναι οι ανάγκες μας εδώ. Και επίσης, μην λησμονούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο ζωτικό για την Ευρώπη. Έναν χώρο που πρέπει να διαφυλάξουμε. Ένα χώρο που τελευταία ανάλυση έχουμε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, να προαγάγουμε, να μην πέσουμε δηλαδή στον αγώνα για την εκβιομηχάνηση παντού και μην ξεχνάμε ότι η γεωργία πάντα θα χρειάζεται επέμβαση, παρέμβαση δηλαδή, στήριξη. Υπάρχουν ε, διάφορες προσπάθειες για διεκδίκηση πόρων για την στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δεν αρκούν όμως αυτά. πρέπει να διατηρηθεί η παρέμβαση γιατί μόνο έτσι μπορεί να διασωθεί η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Φρανκ, πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε στον προπολογισμό πολλές φορές πράγματα που μπορούμε να γράψουμε, να πούμε και κάποια άλλα που μπορεί ή χρειάζεται να γνωρίζουμε συμπληρωματικά. Χωρίς να έχω πρόσθετα στοιχεία αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Ο γεωργικός τομέας κοστίζει 4,2% του ΑΕΠ και είναι περίπου μισό πόντος επί τη 100, 0,5% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν κάνουμε, μια, προσπάθειες για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει και με την ασφάλεια της προμήθειας σε και με το μέλλον της Ευρώπης, ίσως τα ποσά που διατίθενται για τη γεωργία να φανούν κάπως λιγότερο μεγάλα. Δεν ε, προσπαθούμε να σώσουμε μόνο ένα μαγαζάκι που πουλάει τυριά στη τελευταία ανάλυση. Και από το 2012 μέχρι το 2020 θα έχουμε την ε, δέσμευση για διάθεση στα αναπτυσσόμενα κράτη πιο πολλών πόρων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα χρειαστούν. Με τα τωρινά ποσά που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει θα, έχουμε περίπου, θα καλύπτουν περίπου το 1 τρίτο της εκατό, και τα χρήματα δηλαδή. Με επιπτώσεις φυσικά στους ιδίους πόρους. Και αν μιλήσουμε για αφορολόγηση των, ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή των εκπομπών, δίνεται η εντύπωση ότι αυτοί οι νέοι φόροι, εφόσον εγκριθούν, θα εξαντληθούν πολύ γρήγορα, το προϊόν δηλαδή που θα φέρουν, θα εξαντληθεί πολύ γρήγορα ε, εάν δεν αναλάβουμε νέες δεσμεύσεις για την ε, καταπολέμηση των συνεπειών τη χρηματοδότηση κλιματική αλλαγή. Σε μεγάλο περιθώριο χειρισμών δεν έχουμε. Δυστυχώ το διαπραγματευτικό περιθώριο. Περιέγραψε ο Σαλβαδόρ περίπου πόσο θα χρειαστούμε. Περίπου 100 δι ευρώ μέχρι το 2020 για επενδύσει. Αυτό είναι ε, το ποσό μπορούμε να προβλέψουμε μέχρι τώρα. Αλλά Ξέρετε, αυτέ τι μέρε ξέσπασε η μεγάλη κρίση με την Ιαπωνία και τα πυρηνικά και διερωτώμεθα μήπω τυχόν χρειαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθεί πολύ μεγάλη ε, πολύ σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των πυρηνικών στην Ευρώπη και της ε, βελτίωσης των ε, συνθήκων στην πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη πρόκληση για τον προϋπολογισμό και πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες εάν τυχόν είμαστε υποχρεωθούμε κάποια στιγμή στο μέλλον να εγκαταλείψουμε μια τόσο σημαντική πηγή ενέργειας όπως τα πυρηνικά, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά αυτά. Τα λεφτά που έχουμε επενδύσει τα διαγράφουμε. Όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γίνονται καπνός. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και αν μου θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την αναπτυξιακή βοήθεια. 0,7% ο στόχος του 0,7% σημαίνει 30-40 δισεκατομμύρια επιπλέον. Αλλά η τάση είναι ταυτόχρονα ότι όλο και περισσότερη χρηματοδότηση προέρχεται από τον προπολογισμό. Ρωτώ λοιπόν πώ θα το κάνουμε αυτό, χωρί να προσθεθούν και νέοι όροι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τρει νέου τομεί όπου μπορούμε να έχουμε περισσότερο, όπου θα χρειαζόμασταν μάλλον να έχουμε περισσότερο ε, περιθώριο για την αναπτυξιακή βοήθεια και για την ε, αντίδραση σε περιπτώσει φυσικών καταστροφών, είτε εν πάση περιπτώσει ταχεία αντίδραση σε περιπτώσει κρίσεων, αλλά εκεί χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Πρόεδρο, πρέπει να σου <laughs> αφαιρέσω τον λόγο, παρότι με τόση μεγάλη χαρά ακούω τα λουξεμβουριανά γερμανικά σου. Μελωδία για τα αυτιά μου, παρακαλώ. Για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειώσουμε πολύ απλά ότι στον κόσμο ε, έχουμε τεράστιες ε, αλλαγές. Ε, περνάμε στην Ευρώπη από σε μια εποχή που χρειαζόμαστε και ασφάλεια επιστημιστική για τα τρόφιμα, αλλά και ασφάλεια για την παροχή ενέργειας. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική στην Ευρώπη, έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα μας επιτρέψει οικονομικώς καλές εξελίξεις, αλλά παράλληλα και οικολογικές, ε, οικολογική πρόοδο. Και το ένα να μην είναι αντιφατικό με το άλλο, να τα ε, συντονίσουμε. Έχουμε στην γεωργική πολιτική ένα το εξή φαινόμενο. Όλες ε, οι πολιτικές, όλοι οι τίτλοι του προπολογισμού συγκεντρώνονται στην πολιτική αυτή. Θα πρέπει λοιπόν ο προϋπολογισμός ε, να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο όπου, όπου υπάρχουν επικαλύψεις να υπάρχει αποτελεσματικότητα στη χρήση των μέσων και να μην υπάρχει μονομέρεια στην επιβάρυνση. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια γεωργία η οποία θα πρέπει να εντατικοποιηθεί σε κάποιου τομεί, αλλά παράλληλα θα πρέπει να διαμορφωθεί με αποδοτικό τρόπο προκειμένου να μην έχει αρνητικές οικολογικές συνέπειες. Θα πρέπει να δούμε ότι στην Αλία να διασφαλίσουμε ότι και εκεί υπάρχει ε, ε, επιστηστική ασφάλεια, αλλά ότι θα είναι και οικονομική η αλευτική δραστηριότητα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ζημιωθούν τα αλευτικά αποθέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο κλάδος αυτός και Αφενός είναι αντιφατικά τα συμφέροντα αυτά, αλλά αφετέρου το ένα εξαρτάται από το άλλο, γιατί το μόνο ότι είναι οικονομικά αποδοτικό είναι και οικολογικά αποδοτικό σε τελική ανάλυση και αυτό καταδεικνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι περιορισμένος ο προπολογισμό στον τομέα αυτό, γιατί και άλλους ε, τομείς δεν θα μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε αν αποδυναμώσουμε τόσο πολύ αυτό τον βασικό κλάδο. Και αποδοτικότητα τι σημαίνει να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις σε διάφορους τομείς που να λαμβάνουν δηλαδή διπλή χρηματοδότηση. Να πετυχαίνουμε διάφορους στόχους με ένα, ε, με μία γραμμή του προπολογισμού ίσως. Και γι' αυτό θεωρώ ότι στη βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα πρέπει να υπάρχει έλλειψη πόρων και να λάβουμε υπόψη φυσικά και τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρο. λέει η Πρόεδρος, η Ιζαμπέλ Κλείνοντα και μετά ο Σαλμαδόρ. Ευχαριστώ. Ένα πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και νομίζω ότι έχει δίκιο σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να προβούμε σε mainstreaming. Ε, είναι προφανές, αλλά δεν είναι και πνεύμα αυτό. Το mainstreaming θα πρέπει να αποτελεί δεσμευτική προϋπόθεση, διαφορετικά δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί θα γεμίσουμε σε όλες τις σελίδες να φέρουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και παντού θα λέμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, αλλά θα είναι μόνο προθέσεις ε, που θα μείνουν κάστρα στην άμμο. Και ε, νομίζω ότι κάθε φορά που κάνουμε mainstreaming θα πρέπει να υπάρχει μια δεσμευτική προϋπόθεση. Σε ό,τι φορά την αλία, πιστεύω ότι για την αλία πρέπει να λέγουμε λιγότερο αλλά και καλύτερα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εποπτεία και έλεγχος και αν δεν υπάρχει εποπτεία για την υπερελίευση και έλεγχος ε, νομίζω ότι πάλι θα, θα ευωδώσουν οι προσπαθίες μας για τη γεωργία. Είναι ουσιαστικό να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ διατροφής διατήρησης της φύσης κοινωνικού ντάμπινγκ, προστασία των αγροτικών περιοχών και πολλαπλή συμμόρφωση στον πρώτο πυλώνα. Θα πρέπει να υπάρχει πολλαπλή συμμόρφωση στον πρώτο πυλώνα και θα πρέπει να καταργήσουμε τι εξαγωγικέ πιστώσει. Κάρδαλο είναι και αυτό. Τώρα για το θέμα των μεταφορών. Το... Και εδώ έχουμε την εντύπωση, όπως και σε άλλα κεφάλαια, ότι μιλάμε μόνο ε, για τη σημερινή κατάσταση, δεν μιλάω για συνολική αναδιατύπωση, αλλά χρειάζονται κάποιε προσαρμογέ. Τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο διασυνοριακό χαρακτήρα, αλλά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, είναι κάτι που πρέπει να εντάσσονται στους στόχους του 2020. Θα πρέπει να βγάλουμε από την απομόνωση ορισμένες περιοχές και θα δούμε με ποια διατροπικότητα θα το πράξουμε αυτό, δηλαδή ε, να δούμε ποια είναι η προσθεμένη αξία επιτόπου για να έχουμε και ορθές ε, επενδύσεις. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε τις ασυνέπειες και θα πρέπει να μετρήσουμε το θέμα της ε, εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους. Θα πρέπει αυτό να το πράξουμε στις μεταφορές ε, και πρέπει να μειώσουμε τη ζήτηση για τις μεταφορές. Δηλαδή όχι μόνο να διαχειριστούμε τις ροές, αλλά να αποφύγουμε τις άχρηστες μεταφορές και να μειώσουμε τη ζήτηση. Και αυτό μπορεί να γίνει βελτιστοποιώντας ε, τα υφιστάμενα. Θα υποβάλω προς αυτή την κατεύθυνση κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Στην ομάδα που με βοήθησε, η ομάδα που με βοήθησε, αλλά και εγώ προσπαθήσαμε να σεβαστούμε το ρόλο των αντίστοιχων επιτροπών. Δηλαδή αναφέρομαι τόσο και στις ε, επιτροπές που έχουν ε, καταθέσει την αξιολόγησή τους, αλλά και στι επιτροπές που εξακολουθούν να υλοποιούν αυτήν την αξιολόγηση έχουν συνεισφέρει για την εκπόνηση αυτών των διαφορετικών παραγράφων. Εγώ προσπάθησα να μην ε, αναφερθώ εις βάθος στις μεταρρυθμίσεις και στις διάφορες πολιτικές που έχουμε στο κεφάλαιο της αηφορίας, γιατί νομίζω, πιστεύω ότι ε, πρέπει οι αρμόδιες επιτροπές να τοποθετηθούν επί της ουσίας για τη μεταρρύθμιση αυτών των πολιτικών. Εγώ έχω αναφερθεί σε σημείο που έχουμε πολιτική, σαφή πολιτική συνένεση και αυτές οι συνενέσεις φυσικά θα πρέπει να μεταφραστούν και στον προπολογισμό και χρειάζεται φυσικά να λάβει θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού του θέματος, όμως και αυτό είναι επίμαχο για συγκεκριμένες αποφάσεις. Συνειδητοποιώ πλήρως ότι η γεωργική πολιτική η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι βιώσιμη και η αεφορία της ΚΑΠ θα πρέπει να αποκρισταλώνεται και στο πώς συνεισφέρει στο περιβάλλον και στην επιβίωση του τομέα. Δηλαδή η μελλοντική αγροτική πολιτική θα πρέπει να συνδυάζει και τα δύο. Όσοι γνωρίζουν την ΚΑΠ εδώ και πολλά χρόνια θα εκπλαγούν για το πώς η αγροτική πολιτική έχει προσαρμοστεί σε κάποιες ε, μεταβολές και νομίζω ότι αυτό έγινε με απόλυτη επιτυχία. Νομίζω ότι η κοινή αγροτική εκφράζει την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως για να επιβιώσει κάπου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Και επαναλαμβάνω, είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ανακοίνωση του Επιτρόπου Τσόλος και σε ό,τι αφορά το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι για την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 49. Φυσικά η αγροτική πολιτική, όπως και η πολιτική συνοχή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κάποια κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητα αυτά για την προσαρμογή τους στις σημερινές συνθήκες, για την αλία. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις επιδότησης, η Ευρώπη αποτελείται, ξέρετε, από αλείς, από κτηνοτρόφους, από ερευνητές, από ανθρακορίχους κτλ. Και όλοι περιμένουν κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να περισχύουν ε, ε, κάποιοι ε, κλάδι εναντί κάποιων άλλων. Πρέπει να βρούμε λύσεις για όλους και πρέπει φυσικά να αναζητήσουμε και ολοκληρωμένες λύσεις που να μην ζημιώνουν το σύνολο αυτών των κλάδων. Για την κοινή ελευθερική πολιτική πιστεύω ότι έχει πετύχει τους στόχους της που είναι πολλές φορές ταυτόσιμοι με τους στόχους της ΚΑΠ. Είναι σημαντική η επιστημιστική ασφάλεια. Νομίζω ότι η κοινή πολιτική πετυχαίνει του στόχου τη και φυσικά πρέπει να συμπεριληφθούν και περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια εφορία, αν και αυτό πολλέ φορέ θέτει σοβαρά προβλήματα όπω αυτά που ζούμε στην δική μου περιφέρεια τώρα με τι ποσοστώσει. Όμω, όπω και να έχει, μιλάμε για περιβαλλοντικά κριτήρια, κριτήρια εφορία, τα οποία είναι απαραίτητα. Τώρα, για την κλιματική αλλαγή. Φυσικά η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ο πρόεδρος Μπαρόσο μίλησε για τα 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν από την πράσινη οικονομία, 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο σύνολο των 23 εκατομμυρίων ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό αριθμιστικό στοιχείο και έχουμε και άμεσα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας, την εξοικονόμηση καυσίμων και νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις κοινωτικές πολιτικές. Γνωρίζω φυσικά τι σημαίνει αυτό και το υπερασπίζω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον για την ευρωπαϊκή οικονομία δίχω να συμπεριληφθούν τα θέματα τη κλιματική αλλαγή. Αναφέρατε το παράδειγμα τη Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει σε ε, όλα όσα επιδίνωσε στο παρελθόν για να πετύχει την οικονομική της μεγέθυνση. Ε, εδώ ξέρουμε ότι δεν θα θέσει τόσο αυστηρού στόχου όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση με το στόχο αν και άλλες περιοχέ του κόσμου είχαν θετήσει τα ίδια κριτήρια που εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρειάζονταν τώρα να βρισκόμαστε ενώπιος αυτής της επιδείνωσης του περιβάλλοντος ε, ε, που αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι είμαστε σε διαφορετική κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τώρα στην ενέργεια και στα πυρηνικά. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάπως να ηρεμήσουν τα πράγματα για να λάβουμε αποφάσεις ε, για θέματα επενδύσεων στο μέλλον. Εγώ έχω τη δική μου άποψη. Όμω, ε, δεν νομίζω ότι ούτε σε αυτή την επιτροπή στη ΣΟΥΡ, ε, ούτε είναι τώρα η κατάλληλη χρονική στιγμή, ε, ο κατάλληλο τόπο και χρόνο να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων αυτών. Νομίζω ότι η Επιτροπή Ήτρε είναι πλέον αρμόδια για να αξιολογήσει το τι συμβαίνει. Από τη δημοσιονομική σκοπιά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στις διασυνδέσεις, στην καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και στους συνδέσμους που λείπουν στην ενέργεια, στα εφηή δίκτυα. Σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει εξοικονόμηση και αν επενδύσουμε μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση στο μέλλον ε, του κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Εγώ νομίζω ότι αν ε, στοιχηματίσουμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στην ενέργεια και στις μεταφορές ή αν επενδύσουμε στην δημιουργία ενεργειακών δομών σημαίνει ότι στοιχηματίζουμε υπέρ του μέλλοντος και τελικά θα έχουμε πολύ πιο καλά αποτελέσματα και φυσικά νομίζω ότι στην Επιτροπή μας αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ, μάλιστα. Άρα έτσι κλείνει το δεύτερο τμήμα, η δεύτερη φάση της συζήτησής μας και περνάμε τώρα στο τρίτο μέρος, στην συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση να διαβάσω το κατάλογο των ομιλητών. Κωνσταντσε Κρίλ, Ιβα Σκοτμάνη, Γεώργιο Σταυρακάκη, Γιάν Ολμπριχτ, Ντέρεκ Βόν, sofort, äh, José Manuel Fernández, äh, Sidonia Jedrzejewska, ähm, François Alfonsi und Miguel Portas. Okay. Jetzt Konstanze äh, η Κωνσταντσα Κρυλ. Α, συγγνώμη, λάθο. Λάθο, ε, με συγχωρείτε. Ο εισηγητή μα ασφαλώ. Εισαγωγικά να κάνει κάποια σχόλια. Ε, bueno, presento el... Θα σα παρουσιάσω το τρίτο τμήμα που τι τις πολιτικές προτεραιότητες, συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παράγραφη 63 έως 73. Ποιε είναι οι κυρίε ιδέε. Η προστιθεμένη αξία τη πολιτική συνοχή είναι αδιαφεσβήτητη. Πιστεύω ότι ήταν μία από τι ε, πλέον επιτυχεί ευρωπαϊκέ πολιτικέ ε, από τη στιγμή της αναρξής τη, του σχεδιασμού τη. Όμως ε, πρέπει να επισημάνουμε, όπως και είπαμε και για την ΚΑΠ, ότι για να επιβιώσει μία πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται και το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική συνοχή. Πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η συνοχή είναι θεμελιώδης για την επίτευξη στρατηγική Ευρώπη 2020. Όχι μόνο γιατί αν μεταφράσουμε σήμερα στον προϋπολογισμό του 2011 την συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στους διάφορους στόχους της ε, στρατηγικής για το 2020 θα συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική συνοχή ουσιαστικά χρηματοδοτεί όλη την εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020 αλλά και γιατί επιπρόσθετα η πολιτική συνοχή με ένα οριζόντιο χαρακτήρα καλύπτει όλους τους θεμελιώδεις στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την εφόρο ανάπτυξη και την φύη ανάπτυξη. Μια εξυγχρονισμένη πολιτική συνοχής και μια ισχυρή πολιτική χρειάζεται παρκή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ό,τι έχουμε στις σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι υπάρχει και γενική συνένεση τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ από τις συζητήσεις που είχαμε σε αυτή την Επιτροπή ΣΟΥΡ και από τις εκθέσεις της ε, Επιτροπής για την Περιφερειακή Πολιτική. Δεν πιστεύω ότι κάνει επιζητά μείωση των πόρων για την πολιτική συνοχή. Μιλάμε απλώ για προσαρμογή. Όπως και να έχει, η πολιτική συνοχή πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα πλέον προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από το σημερινό earmarking, από τη σημερινή ε, ενεργοποίηση των πόρων. Αυτό πιστεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτές οι συμβάσεις που πρέπει να γίνουν μεταξύ κομισιών, κρατών μελών και τοπικής αυτοδιοίκησης Νομίζω ότι καθυστερεί πολύ η Κομισιόν στο να προσδιορίσει τις συμβάσεις αυτές και τελικά αυτό προκαλεί αβεβαιότητα σε όλο τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και νομίζω, όπως και να έχετε, οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία περνά από την ε, σύσταση αυτών των συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Εδώ Πρέπει να υπάρχει και συσχετισμό με τα διάφορα διευθυντικά ταμεία. Γι' αυτό μιλάμε για ένα διαφορετικό επιτομέα. Μιλάμε για την αστική διάσταση. Ότι πρέπει η διάσταση αυτή να συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική συνοχή. Και κάτι ακόμη σημαντικό που ήταν και στόχος των τελευταίων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης ως ποιο βαθμό η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνδέεται με κριτήρια μακροοικονομικής πολλαπλή συμμόρφωσης. Εγώ εδώ έλαβα τη θέση ότι δεν πρέπει να συνδέεται γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια στρεβλά αποτελέσματα. Δηλαδή να έχουμε εθνικές οικονομίες ε, που απομακρύ, αυτές οι οικονομίες που απομακρύνονται από τα πρότυπα της οικονομικής διακυβέρνησης αν ε, τις τιμωρήσουμε ακόμη περισσότερο τελικά τι θα κάναμε θα επιδεινώναμε τα προβλήματα αυτών των οικονομιών αν στερούσαμε δηλαδή και τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής είναι μια ιδέα που αναφέρω εγώ στην εκθεσή μου το υπερασπίστηκα και στην πολιτική περιφερειακή συνοχή, ελπίζω να διατηρήσουν την ιδέα αυτή οι συνάδελφοι. Αυτά για την πολιτική συνοχή, Πρόεδρε. Και τώρα η Κωνσταντζα Κρυόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή, γιατί θεωρώ ότι αυτά που γράφει για την ε, πολιτική συνοχή στην έκθεσή του αποτυπώνουν τις σημαντικότερες προτεραιότητες τις οποίες συζητήσαμε στην Επιτροπή Ρέγγι. Και αυτό φυσικά το υποστήριξε και η ομάδα μου. Ωστόσο, παρόλα αυτά θα ήθελα σε κάποιες κατευθύνσεις να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην έκθεση. Θεωρώ ότι η πολιτική συνοχή ε, είναι η κατάλληλη και στις διαπραγματεύσεις ε, του μελλοντικού προϋπολογισμού στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θετική βάση διαπραγμάτευσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δοθεί έμφαση στα key priorities, στις βασικές προτεραιότητες, ότι είναι σημαντικό για όλους τους στόχους τους οποίους ε, προασπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται διαφορά, να διαφορές μεταξύ των ε, περιφερειών. Αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές. Και ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην πολιτική συνοχή, προκειμένου να καταστεί και πιο διακριτή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το ενισχύσω αυτό περισσότερο για να έχουμε καλύτερη την πραγματευτική θέση με την συνθήκη της Λισαβόνας. Η εδαφική συνοχή ε, είχε τονιστεί εκ νέου, γιατί υπήρχε πάντα τέτοια πολιτική συνοχής, αλλά δόθηκε νέα έμφαση και αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε. Στο κεφάλαιο τώρα για την πολιτική συνοχή θεωρώ ότι θα πρέπει να διασαφινιστεί ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει και μπορεί να ε, αξιοποιηθεί από όλες τις περιφέρειες, από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί αυτό το επιχείρημα του, των καθαρών ε, εισφορέων και των καθαρών ε, αποδεκτών ε, μπορούμε να το αποδυναμώσουμε έτσι. Τώρα, μία παρατήρηση για τις αρνητικές προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή πρέπει να πω το εξή ότι δεν ζητάμε πιο πολλά, αλλά δεν θέλουμε και λιγότερα από αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας μέχρι τώρα. Αλλά απαιτώντα αυτό, τι σημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εξυγχρονιστεί με τέτοιο τρόπο και να γίνουν ε, κατά τόπους ε, αποταμιεύσεις οικονομίες προκειμένου αυτά που έχουμε στην πολιτική συνοχή να ληφθούν πιο πολύ υπόψη σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος, της δημοκρατικών ε, εξελίξεων, θέματα εδαφικά, ενίσχυση της έρευνας που διατίθεται, την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν εμεί να κάνουμε οικονομία. Το αντίθετο, μάλλον ε, χρειαζόμαστε πιο πολλά. Θα μπορούσαμε να, να απαιτήσουμε πιο πολλά κονδύλια, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ πειθαρχημένοι. Ο κ. Κουτμάνη. Ευχαριστώ. Καταρχά, θα πρέπει να πω είναι ότι το κείμενο εδώ πέρα για την πολιτική συνοχή ε, είναι πάρα πολύ πλούσιο. Είναι πολύ πιο πολλά διπλάσια στον αριθμό τα κεφάλαια που αναφέρονται από τη για τη Γεωργία, αλλά τα πράγματα με τη χρηματοδότηση είναι αντίστροφα. Να πω στο 66 το εξή. Πιστεύουμε ότι αυτή η νέα ε, συμφωνία εταιρική σχέση θα περιλαμβάνει, και αυτό αναφέρθηκε και στην έκθεση Βάκνερ, όπου είπαν ότι κάθε τρία χρόνια θα ε, υπάρχει ανάλυση αποδοτικότητας απορρόφησης των κονδυλίων. Πιστεύουμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμπεριληφθεί αυτό. Κατά δεύτερον, στο 69 δεν θα υποστηρίξω το 69, γιατί εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, μιλάμε για απλοποίηση. Αλλά εμένα μου φαίνεται φιλοσοφικό το ζήτημα αυτό. Γιατί η Επιτροπή, δημιουργώντας ε, ένα σύστημα χείριση τριών επιπόδων, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των μεγάλων project, έχει πετύχει να περιοριστεί ο ρυθμός των σφαλμάτων και των απάτων πολύ σημαντικά. Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να κάνουμε περαιτέρω απλοποίηση, γιατί οι χώρες έχουν αποδεκτικά στοιχεία και αυτό τι σημαίνει ότι μπορεί το σύστημα να είναι αποδοτικό. Κάθε περαιτέρω απλοποίηση, απλούστευση δεν θα είναι παραγωγική, γιατί θα αυξηθούν ενδεχομένω οι απάτες ή, εν πάση περιπτώσει, οι κακο η κακή χρήση των πόρων. Στο 71 τέλος. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόταση, γιατί κανονικά μιλάμε για το 4% του ΑΕΠ, το ποσοστό των ιδιωτικών ταμείων. Καταλαβαίνω ότι αν θέλετε να αποβεί αυτό εις βάρος της πολιτικής συνοχής. Ίσως όμως θα έπρεπε να το γράψουμε λίγο πιο καθαρά. Πρόκειται για λεφτά που προορίζονται για σχέδια και αν θέλουμε να παραμείνουμε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και τηρώντας το 3% δεν θα γίνει αυτό ε, εις βάρος ε, της ε, συνοχής να γράψουμε συγκριματοδότηση. αν αυτό εννοείται, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Και τώρα Γιώργιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, από πλευράς μου θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση, είναι καλή και αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα εργαστούμε στο μέλλον. Πιστεύω επίσης ότι η παρουσία, ο έντονος ρόλος της ε, πολιτικής συνοχής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει τονιστεί επαρκώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια θέματα της έκθεσης, επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο λογικό να υπάρχει υποκεφαλίδα για την ε, συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση μετά την γνώση και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θεωρώ επίσης ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, ε, από το στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την, ε, τα αποτελέσματα, την καταβολή των δαπανών και τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να πω και εγώ ότι η έκθεση και σε αυτό το σημείο είναι πολύ καλά διατυπωμένη. Θα ήθελα μόνο κάποια σημεία να επισημάνω. όπου νομίζω ότι η συμπληρωματικότητα με άλλα κομμάτια της εκθέσεως θα μπορούσε να βοηθήσει. Εκεί που γίνεται λόγος για νέες προκλήσεις, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι μεγάλη πρόκληση είναι οι ανισότητες. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι όταν μιλούμε για έρευνα, ανάπτυξη και ερωτομία, πάλι σημειώνονται δυστυχώς ανισότητες, τις οποίες θα μπορούσαμε να μετριάσουμε χάρη σε μια καλή πολιτική της συνοχής τα μέσα της οποίας, τα κονδύλια της οποίας θα πρέπει πρωταρχικά να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται και σε άλλα σημεία της έκθεσης. Είναι σημαντικό λοιπόν, πέραν των λοιπόν ταμείων, αναφέρονται και το, αναφέρονται και το Ταμείο Συνοχής. Και θα ήθελα να διατυπώσω το εξή ως ερώτημα. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε σαφές ότι χρειάζεται να έχουμε βελτίωση και της ε, διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ερώτημα επίσης ανοιχτό. Στην πολιτική της συνοχής συζητήθηκε στο Συμβούλιο όχι η στήριξη της πολιτικής συνοχής, αλλά η οπισθοδρόμηση στο multi-finance systeming, δηλαδή στα πολλαπλά ταμεία, οι πολλαπλά συστήματα χρηματοδότησης. Πρέπει όντω να επιστρέψουμε σε αυτό το σύστημα. Θα είναι καλύτερη έτσι η πολιτική συνοχή, μια και αποδεικνύεται ότι δεν έχει λειτουργήσει μέχρι, καλά, τώρα αποτελεσματικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βον θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο τμήμα αυτό της έκθεσης, το οποίο μου φαίνεται κάπως πιο λεπτομερές από τα άλλα τμήματα. προτεραιότητα μα για τι προσεχεί δημοσιονομικέ προοπτικέ όντω θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε να τη στηρίξουμε αυτέ τι εργασίε και την απασχόληση, βεβαίω χρειαζόμαστε την πολιτική τη συνοχή. Στην παράγραφο 65 όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα χρηματοδότηση τη τρέχουσα περίοδου στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Δεν ξέρω αν εννοεί πραγματικού όρου, ποσά δηλαδή, ή ποσοστό επί του ε, προπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα για την πολιτική συνοχή. Και εν γέννη, συμφωνώ με το πνεύμα τη ε, παραγράφου 65. Στην παραγράφου 66 αστικά κέντρα πόλης. Βεβαίως, ξέρουμε όλοι ότι είναι κινητήρη μοχλή στην οικονομική δραστηριότητα. Και πάντοτε όταν ακούμε και τους εκπροσώπου τη να μιλάνε, υπογραμμίζουν τη σημασία των αστικών κέντρων και των πόλεων. Αλλά θα ήθελα να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί στη διατύπωση του τι σημαίνει φερειπίνα αστική διάσταση και πόλη. Διότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη ή οι περιφέρειες οι ίδιες να επιλέξουν τον ορισμό αυτών του αστικού κέντρου. Επίσης παραπέρα ε, όπου γίνεται λόγος για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην παράγραφο 71 ε, ε, υπόθηκε από κάποιους ότι θα πρέπει να συνδεθεί με τη συνοχή. Ε, όμως το να πούμε σε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα οικονομικά ε, ότι σκοπεύουμε να τους ζητήσουμε περισσότερα χρήματα τα οποία θα πάνε στη χρηματοδότηση θέσεων εργασία και απασχόλησης πάλι στα ίδια τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι είναι παλαβομάρα, λέει ο μιλητή, και ίσως θα πρέπει να το διαγράψουμε. Και εν τέλει, μια γενική παρατήρηση. Το συνολικό ποσό που θα εγγραφή στις ερωτικές δημοσιονομικές προοπτικέ μετά το 2013. Πρώτα πρέπει να το γνωρίζουμε και μετά να προσδορίσουμε την ε, κατανομή των ποσών στι κύριε προτεραιότητες. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή χρηματοδότηση λοιπόν. Και μετά να ξέρουμε, εξαίροντας τα ποσά, να προσδορίσουμε τις προτεραιότητες μας. Ευχαριστώ. Ζωζέ Μανουέλ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και επίσης συμφωνώ ότι η πολιτική συνοχή ε, αυτή η καθεαυτή μεταφράζει την προσθεμένη αξία που όλοι γνωρίζουμε. Φυσικά όλες οι χώρες ε, επωφελούνται από την πολιτική συνοχή ε, και ακόμη και αυτές που λαμβάνουν περισσότερα βοηθούν ε, τελικά όσους λαμβάνουν λιγότερο και όλοι κερδίζουν με αυτή την πολιτική συνοχή όπως φαίνεται από μια σειρά Η πολιτική συνοχή έχει περισσότερη ζωή και ξεπερνάει τη στρατηγική για το 2020 είναι ανεξάρτητη από τη στρατηγική αυτή. Σε ό,τι αφορά το σημείο 66, Λέει ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητες. Εγώ θέλω να αναφερθώ αν ε, εδώ η αηφόρος ανάπτυξη και η καθολική ανάπτυξη ε, πρέπει να συνάδουν με την πολιτική συνοχής. Ε, αυτό εννοείται Ίσως θα ήταν πιο σωστό να πούμε ότι υπερασπίζουμε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 θα πρέπει να συμφωνεί με τους στόχους με τους πέντε στόχους που έχουμε στη στρατηγική για το 2020 η πολιτική συνοχής είναι δυνατό να πλουστευτεί, είναι δυνατόν να προσανατολιστεί προς μια πολιτική αποτελεσμάτων. Επίσης, ε, είναι δυνατόν ε, να δώσουμε και ιδιαίτερη έμφαση σε όσους παράγοντες την προωθούν. Και σε αυτό που υπάρχει στο 65, για την προσέγγιση εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση ότι δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το σημερινό δημοσιονομικό προγραμματισμό. Σε αυτό συμφωνώ. Και μάλιστα θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε και για κάποια ποσοστία αύξηση. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, αλλά και ο κάθε πολίτης, τι συμβαίνει με αυτά τα χρήματα είναι πολύ εύκολα, πολύ εύκολο παραδείγματο χάρη να δημοσιεύονται όχι μόνο τα προγράμματα που είναι υπό εκτέλεση, αλλά και τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί. Είναι ένας τρόπος ε, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε μια ευρύτερη περιοχή, γιατί υπάρχουν ε, χώρες ε, όπως η δική μου ε, που ε, βρίσκονται σε διαφορετικές κατηγορίες και δεν λαμβάνουν όλες οι περιοχές τα ίδια κονδύλια. Η συντονισμός με το ΕΚΠΑ είναι σημαντικός. Όμως, για μένα το κατακεφαλήν ε, θα πρέπει να διατηρηθεί με το κύριο κριτήριο. Υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που έχει να κάνει με τις ενδιάμεσες περιφέρειες ή με τις ε, ε, phasing out περιφέρειες ε, σε μεταβατικό στάδιο. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε το καθεστώς phasing out και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοεί η Επιτροπή όταν αναφέρεται σε ενδιάμεσες περιφέρειες. Ευχαριστώ και νομίζω ότι φυσικά ότι είτε μιλάμε για τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της πολιτικής συνοχής, ένα είναι σαφές ότι δεν... Ε, δεν κρατίζουμε εδώ την νομοθεσία η οποία θα ακολουθήσει μετά βάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτώντας τις λεπτομέρειες ε, των ζητημάτων αυτών. Η Σιδονία τώρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεται διεξοδικά στην έκθεση, στην Πολιτική συνοχή του σχέδιου εκθέσεως, αλλά θα ήθελα, και αυτό είναι πολύ καλό, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις μάλλον γενικότερες. Καταρχάς, θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η πολιτική συνοχή. δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον αντίον, η πολιτική συνοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με, την ίδια, με τα ίδια τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλάμε για τις βασικές ελευθερίες, την ιστορική αγορά, που έχει πολύ ε, στενή σχέση με την ε, πολιτική συνοχή. Οι τέσσερις ελευθερίες λοιπόν, διακίνησης εμπορευμάτων υπηρεσιών, προσώπων, είναι προϋπόθεση απαραίτητη για την ουσιαστική λειτουργία της πολιτικής συνοχής. Για να αποβεί αυτή επωφελής και βέβαια για τους αποδέκτες της, αλλά και για να λειτουργήσει ολόκληρη, ολόκληρο το δόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ακριβώς βλέπω να μην γίνεται επαρκής συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχής συχνά δυστυχώς ε, αντιμετωπίζεται ως μια μεταφορά πόρων από τους πλούσιους προς τους φτωχότερους. Δεν είναι αυτό όμως, γιατί όλοι υποφέρουν από μια καλή πολιτική συνοχή. Ανυψώνονται βέβαια οι φτωχότερες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως με αυτό είναι σε θέση να διαθέτουν και προσφέρουν πόρους και ενδεχομένως να αυξήσουν την εντό αγωγικών καταναλωτική τους δυνατότητα, δηλαδή να αξιοποιήσουν περισσότερους πόρους και τεχνολογίες. Αυτό είναι προ τον των πάντων. Βελτιώνονται επίση οι εξαγωγικέ δυνατότητες για όλους. Και μην ξεχνάμε ότι η πολιτική συνοχή είναι εκείνη η οποία εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, των ελευθεριών πάνω στου οποίε στηρίζεται η εσωτερική αγορά. Και έχω ακόμα μια παρατήρηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές πιέσεις, έντονες πιέσεις, γίνεται λόγος για μείωση του κόστους, περιορισμό των ποσών κτλ. Φυσικά προσπαθούμε με τα χρήματα που έχουμε στη θέσή μας να εξασφαλίσουμε ως το δυνατόν πιο καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Εγώ ξέρετε ότι έχω αυτή την ε, μονομανία της πολιτικής για την νεολαία, για τους νέους. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν κοστίζει τόσα λεφτά. Έχουμε το πρόγραμμα Youth in Action, παραδείγματο χάρη, το οποίο επιτρέπει στους νέους μας να προετοιμαστούν πιο ουσιαστικά, πιο καλά για την αγορά εργασίας που είναι 50 φορές πιο φθηνό από άλλα προγράμματα που έχουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Βεβαίω, δίκιο έχετε και από την άλλη, η πολιτική συνοχή έχει φέρει καρπού όχι μόνο όταν έχουν φέρει πλούσιοι, όταν έχει φέρει τι φτωχότερε περιοχέ σε επίπεδο τέτοιο ώστε να φτάσουν στο επίπεδο πλούτου των πλουσιότερων περιοχών, αλλά ήδη από τη στιγμή που αρχίζει να τι ε, στηρίζει τι φτωχότερε ε, περιοχέ, φέρνει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό το είχαμε σαν ε, ε, κραυγαλαίο παράδειγμα με την ε, κατασκευή αεροδρομίων Φερρυπίν στι ανατολικέ περιοχέ τη Γερμανία, που αμέσω αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα μα. Την υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα πρέπει να αναλάβουμε ουσιαστική δράση και να κινητοποιηθούμε, διότι ενδέχεται η πολιτική συνοχή να είναι η αρνητική ε, προτεραιότητα στον προπολογισμό. Δηλαδή αυτή η κατηγορία ε, πολιτικής που θα μείνει τελευταία στη χρηματοδότηση και όχι πρώτη. Ε, πρέπει λοιπόν να προαγάγουμε τις πολιτικές μας εκείνες οι οποίες προσφέρουν προσθεμένη αξία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Δεν στηρίζει μόνο τις πιο φτωχές περιοχές και αυτές που, στις οποίες πηγαίνουν τα χρήματα αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό Ορίζουμε λοιπόν εδώ και καιρό μια πολιτική συνοχή. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει καταλήξει σε, στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ότι η Ευρώπη δεν έχει την απαιτούμενη συνοχή. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική συνοχή. Και επιπλέον θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν πρόκειται πάντα για, πολιτι... για περιοχέ οι οποίε έχουν έχουν πίσω του το βαρύ παρελθόν του σιδηρού παραπετάσματο και όλα ο Νόη έχει, έχει φέρει στην ιστορία αυτών των κρατών το σιδηρού παραπέτασμα, αλλά και άλλες περιοχές. Μην κλείσουμε ότι υπάρχει μεγάλη κρίση. Σήμερα, αύριο, η ελληνικέ περιφέρειε, Ιρλανδικέ, ξέρουμε πώ θα βγουν από την κρίση. Μπορούν να βγουν αλόβητε. Ναι, αλλά μόνο χάρη στην πολιτική συνοχή. Ε, δηλαδή, αν αυτή η πολιτική συνοχή καταστεί ένα διαρκέ εργαλείο τη ευρωπαϊκή πολιτική, με μια ρύθμιση τακτική της εδαφικής συνοχής, όπως ζητάμε και στη δημοσιονομική συνοχή και λειτουργία. Δηλαδή, η πολιτική συνοχής μπορεί να εξασφαλίσει πιστώσεις οι οποίες σήμερα χορηγούνται για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χρειαστεί να πολλαπλασιάζονται στο μέλλον προκειμένου να λύσουμε προβλήματα των υπερπληθών ε, αστικών κέντρων ή της ε, περιμομένης υπαίθρου, αλλά να έχουν εξασφαλίσει αυτή την ισορροπία εγκαίρως. Αυτά λοιπόν και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε και μια οικονομική χρηματοδότηση και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε ιδιαίτερα την έννοια της ενδιάμεσης περιφέρειας η οποία επιτρέπει την οργάνωση της περιφερειακής πολιτικής μακροπρόθεσμα και ταυτόχρονα να ξεπεράσουμε την αυστηρή θεώρηση που είχαμε πριν από 7 χρόνια ε, μια πολύ στενή θεώρηση δηλαδή, εν ώψη βέβαια και της εντάξεως των νέων κρατών μελών. Μια γενικότερη θεώρηση λοιπόν λέγω είναι ο καλύτερος τρόπος να αποτελέσει μια βιώσιμη πολιτική και να φέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα η πολιτική συνοχής. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση βλέπω ότι δεν έχουν ε, ενσωματωθεί στις προτάσεις του συγκεκριτού οι διασυνοριακές δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτές βοηθούν χώρες τις οποίες είχαμε ξεχάσει επί δεκαετίες, τις οποίες είχαμε στρέψει, είχαμε στρέψει από την πλάτη εδώ και δεκαετίες και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αναπτύξει αυτές τις μακροπεριφέρειες, τις διασυνοριακές συνεργασίες, μπορούμε να ε, περιμένουμε σαφή ζήτηση από αυτές τις περιφέρειες και άρα θα πρέπει να τις ενισχύσουμε στο πρόγραμμά μας. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει ο εισηγητής να δώσει πιο πολύ έμφαση στο κοινό πλαίσιο στρατηγικής, να είναι πιο θαραλέος ενδεχομένω και στα δημοσιονομικά μέσα, δηλαδή το 1973. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Πόρτας. Ευχαριστώ να ξεκινήσω από το εξή. Συμφωνώ με το σημείο 71 της ε, πρότασης της έκθεσης και γενικά συμφωνώ με όλες τις παραγράφους που αναφέρονται στην απλουστεύση των διαδικασιών, στην αξιολόγηση βάση αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν δηλώνω τη συμφωνία μου. Επίσης συμφωνώ με την πρόταση του συναδέλφου Αλφορσή για το να εξετάσουμε την, ε, το καθεστώς της ε, ενδιάμεσης περιοχής μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τώρα, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που μας τίθεται στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, ο συνάδελφο ε, έχει δίκιο όταν είπε ότι οι περιφερειακέ χώρες που βρίσκονται δυσκολίε ε, θα ήταν πολύ χειρότερα σήμερα δίχω την πολιτική συνοχή. Επίση, είναι αλήθεια ότι οι συνοχής συνοχή ε, ήταν ανεπαρκείς. τελικά, αποκαλύφθηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης των διαστάσεων που βιώνουμε. Έτσι λοιπόν και τα δύο αυτά είναι αληθή και εμείς ε, δεν πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε ε, εθνικοποιημένα ευρωπαϊκά κονδύλια, αν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε ένα εργαλείο πολιτικής καθαρά ευρωπαϊκό. Δηλαδή ε, αυτό ε, πρέπει να απαντά σε προτάσεις που γίνονται από το κράτος, δηλαδή υπάρχει σε χρηματοδότηση. Η δική μου αμφιβολία είναι αν χρειαζόμαστε ακριβώς ένα ταμείο το οποίο για θέματα φτώχειας και κοινωνικής σύγκλησης Ε, που να μην έχει καθαρά χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητα. Δηλαδή τι εννοώ, θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Αυτή η κρίση είχε ως ε, αποτέλεσμα τα συντοξιδοτικά συστήματα στις περιφερειακέ χώρες να παγώσουν ή μάλιστα να μειωθούν και οι συντάξεις σε πολλές περιπτώσεις. Τα συστήματα κοινωνική στήριξη. Δεν συμβαίνει το ίδιο στι πλούσιε χώρες. Δηλαδή η κρίση στο στρατηγικό πλαίσιο ε, αποκλήσεων μάλλον παρουσιάζει αποκλήσεις μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών και η κρίση οδηγεί στο να αυξηθούν οι ανισότητες όχι μόνο στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Δηλαδή αυξάνονται ε, και μεταξύ των χωρών γιατί αυξάνεται η απόκληση μεταξύ των χωρών. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα εργαλείο, ένα μέσο συμπληρωματικό έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντισταθμίσει την αύξηση των αποκλήσεων σε ό,τι αφορά την επιδείνωση της φτώχειας ή της επιδείνωσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Και η χρηματοδότηση δεν θα γίνει από τους πόρους που έχουμε σήμερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, όμως αυτό το πρόβλημα είναι στρατηγικό πρόβλημα. Αν θέλουμε να επερασπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικής Σύγκλησης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τσέλερ, τελευταίο ομιλητή. Και ο Σαλβαδόρ για να κλείσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ από πλευρά μου τον εισήγητη, τον κύριο Καρικαπογέδο, που έλαβε στο μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη την ε, γνωμοδότηση τη επιτροπή περιφερειακή πολιτική στην έκθεσή του. Με χαρά βλέπω ότι είναι πολλοί οι συνάδελφοι οι οποίοι υποστηρίζουν την πολιτική συνοχή. Ακριβώς η πολιτική συνοχή είναι εκείνη η οποία ιδιαίτερα μετά την τελευταία, τις τελευταίες διευρύνσεις μπορεί να διαφυλάξει την σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Επιτρο... Ε, και μάλιστα αποδεδειγμένα. Και εφόσον είναι έτσι, στο πλαίσιο και των δομών και του δημοσιονομικού προγραμματισμού πρέπει αυτό τον όρο να τον λάβουμε υπόψη, τη σημασία δηλαδή, της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ τις ε, κυρίες Φερνάντες και η για, για τα όσα είπαν. Θα υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια πολιτική η οποία δεν έχει μόνο αμυντικό χαρακτήρα, αλλά διαρθρωτικό. Το είδαμε άλλωστε στη συζήτηση του τελευταίου μήνε ότι ο καθένα προσπαθεί από το δικό του τομέα και για λογαριασμό του να εξασφαλίσει το δυνατόν πιο πολλά χρήματα για συγκεκριμένα έργα, ε, και είναι μια συζήτηση αυτή την οποία έχουμε πραγματοποιήσει και σε επίπεδο των επιμέρου επιτροπών του Κοινοβουλίου. Προσπαθεί δηλαδή ο καθένα για, για το δικό του πολιτικό τομέα να εξασφαλίσει πιο πολύ χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν έχει η πολιτική συνοχή πολύ μεγάλη σημασία γιατί καλύπτει διάφορους τομείς ε, πολιτικής και βλέπω δυστυχώς απόκληση σε σχέση με τις προτινόμενες δομές των μεσοπρόθεσμων, του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα στο σημείο 1 με την αναφορά στην πολιτική, τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, όπου ορίζονται οι δομές. Και μετά έχουμε στο 1α ανάπτυξη, απασχόληση, β, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, γ, πάλι ανάπτυξη για την απασχόληση και μετά μόνο έρχεται η πολιτική συνοχή. Αυτό τι σημαίνει, ότι εάν όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή, δηλαδή κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Μεταφορών, δηλαδή διαρθρωτική πολιτική, στο 1α και το 1β, εάν τα αναφέραμε όλα αυτά, ως αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, δηλαδή την κλαδική κατανομή, την τομεακή κατανομή της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη και γενικότερη θεώρηση, έτσι ώστε να έχουμε τα λειτουργικά μας προγράμματα για τη μεσοπρόθεσμη πολιτική, όπως θα θέλαμε. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 αποτελεί βέβαια ένα όρο και προσδιορίζει το περιεχόμενο των πολιτικών μας με ορίζοντα το 2020. Αλλά μην γελιόμαστε, έξω από το Κοινοβούλιο δεν απασχολεί κανέναν αυτή η, πολιτική, αυτή η στρατηγική για το 2020. Και η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών των εθνικών κρατών πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και αν θέλουμε να την φέρουμε σε αίσιο πέρας θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις υφιστάμενες δομές, αυτές που έχουν αποδείξει την αξία τους. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Όσον αφορά τη δομή και τη διάρθρωση του προπολογισμού, ο εισηγητή ακολουθεί την υφιστάμενη δομή όπως βλέπετε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν και παρακαλώ να μην μιλάμε με υποσημειώσεις και λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι, να κοιτάμε τους βασικούς στόχους. Τις λεπτομέρειες τις βλέπουμε το απόγευμα. Ε, και τώρα παρακαλώ το Σαλβαδόρ να λάβει το λόγο για να καλύψει και το, την αυτή, το τρίτο σημείο τη της δεύτερης αυτής φάσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, καθώς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ε, δεν ε, θέλησα και εγώ να μπω σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Βέβαια, συμφωνώ με τη θέση της Επιτροπής Ρέγκη. Νομίζω ότι όσα υπόθηκαν και στις συνενέσεις τις οποίες κατέληξαν ε, στην αρμόδια επιτροπή, ε, εγώ τις έχω αντικατοπτρίσει εδώ. Τώρα, για μένα η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν είναι ένας ε, στόχος, αλλά ένας δρόμος, μία οδός. Μας δείχνει η στρατηγική Ευρώπη 2020 πώς θα βελτιώσουμε τις κοινοτικές δαπάνες για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι η στρατηγική για το 2020 συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινοτικές πολιτικές και πολύ συγκεκριμένα την πολιτική συνοχής. Δίχως πολιτική συνοχής, μικρινά, πάρα πολλά κράτη-μέλη θεωρώ ότι δεν θα ήταν σε θέση να αντισταθούν στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση ε, που βιώνουμε από το 2008 έτσι λοιπόν θεωρώ ότι οι πολιτικές συνοχής ε, πρέπει να είναι για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το κράτος τους ή την περιφερειά τους. Και τις προάλλες, το αναφέρα γι' αυτό σε μια συζήτηση, υπάρχουν και περιοχές στη Βόρεια Σουηδία για τις οποίες χρειάζεται πολιτική συνοχής όπως ε, και οι πολίτες της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να έχουμε μια πιο καθολική εστίαση στην πολιτική συνοχή. Πιστεύω ότι σε αυτό όλοι συμφωνούν. Τώρα, η προσαρμογή της πολιτικής συνοχή, Ο όρος προσαρμογή είναι ορό κλειδί. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικές αυτές οι αναπτυξιακέ συμβάσει που θα πρέπει να συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κάθε τομέα. Μέχρι να έχουμε επιτάπητος ε, πιο συγκεκριμένα στοιχεία για αυτές τις συμβάσεις, θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε κριτήριο πολλαπλής συμμόρφωσης για τα διαφορετικά ταμεία. Εγώ συνεχίζω εδώ να περιμένω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ε, και αυτά τα δικατοτρίζω σε κάποια από τις παραγράφους της έκθεσης, απλούστευση. Πιστεύω ότι η απλούστευση είναι απαραίτητη πλούστευση δεν σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο έλεγχο σε καμία περίπτωση. Και αν ε, θεωρήσουμε ότι η απλούστευση σημαίνει λιγότερο έλεγχο, τότε εγώ απέτυχα στη σύνταξη του εδαφείου 71. Νομίζω ότι η απλούστευση διευκολύνει τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης Έχουμε τελικά λιγότερα λάθη και σεβόμαστε και αυτό που, ζήτησε πάντοτε, που ζητά πάντοτε η Επιτροπή του Ελέγχου του Προπολογισμού για το θέμα των διαθέσιμων πόρων. Είναι μια έννοια που δεν ήθελα να συμπεριλάβω στο κείμενο, αλλά που υπάρχει όμως ε, στις ε, ανησυχίες των μελών της Επιτροπής ΡΕΙΚΙ, είναι το εισόδημα της συνοχής. Δηλαδή είναι προφανές ότι θα υπάρχουν λιγότερες περιοχές που θα είναι στο στόχο σύγκλησης από το 2014 και μετά. Ακόμη και αν η οικονομική κρίση παρουσιάζει, επιφέρει παράδοξα αποτελέσματα. Δηλαδή οι περιφέρειες που ήδη ήταν στο στόχο της ανταγωνιστικότητας ίσως ε, φέτος να είναι σε κατάσταση phasing in. Και όσες ήταν σε phasing in σε αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, τώρα να βρίσκονται σε στάδιο phasing out. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιες θα είναι οι περιφέρειες που θα συνεχίζουν να είναι στο στόχο σύγκλησης. Γιατί μέσα από αυτό το εισόδημα συνοχής ε, εκεί μπορούμε να επικεντρωθούμε στα όσα ανέφερε ο κ. Φερνάντες στις ε, περιφερειές που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση. Και δεν ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ, ούτε κι εγώ να τοποθετηθώ επ' αυτόν, γιατί όπως σας είπα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και προτιμώ λοιπόν να έχω μια πιο γενική θεώρηση για το τι είναι απαραίτητο σε μια πολιτική συνοχή. Δεν προτίμησα να μπω σε λεπτομέρειες, ούτε επί των κριτηρίων, ούτε επί των περιφερειών που θα έπρεπε να εντάσσονται στους διάφορους στόχους. Αυτό θα γίνει σε μια μετέπειτα φάση, σε ένα μετέπειτα στάδιο της έκθεσης. Όμως για την πολιτική συνοχή είτε μιλάμε για ποσοστά είτε για καθολικά ποσά δεν μπορούν αυτά να βρίσκονται κάτω των σημερινών επιπέδων αν θέλουμε τελικά να πετύχουμε όλους τους στόχους. Η επέκταση της πολιτικής συνοχής στις ιδιαιτερότητες της κάθε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, θα πρέπει να λάβει χώρα και επίση θα πρέπει να πληρούνται και προποθέσει χρηματοδότηση των υποδομών, των νέων προτεραιοτήτων ε, που θέτει η Στρατική Ευρώπη 2020. Ε, Συνάδελφος ε, έχει δίκιο, εγώ φταίω. Δεν συμπεριέλαβα το θέμα της σύγκλησης όπως μου είχαν προτείνει. Ε, δεν το συμπεριέλαβα στις προκλήσεις, ελπίζω να γίνει μέσω τροπολογιών. Κοιτάξτε, όταν έχουμε τόσο μεγάλες εκθέσεις, ε, πολλές φορές την χάνει να ξεχάσουμε και να συμπεριλάβουμε ορισμένες προτάσεις. Ε, όταν είχα λάβει την πρόταση αυτή μου φαινόταν πολύ καλή. Λυπάμαι, λυπάμαι που δεν το συμπεριέλαβα στην έκθεση, αλλά προλαβαίνουμε ακόμα. Μιλούσαμε για το σημείο 65, για την ε, συμπερίληψη ποσοστών αριθμητικών στοιχείων. Δεν θα γίνει αυτή η συζήτηση τώρα, αλλά στο μέλλον. Χρειαζόμαστε απλώς επαρκή χρηματοδότηση, αυτό αναφέρω εδώ και για το 71 για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Η πολιτική συνοχή δεν πρέπει να πληρώνει δις τα λάθη των κρατών μελών που δεν μπόρεσαν να σεβαστούν τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και τους στόχους σύγκλησης για την παρουσίαση και τη δομή. Θα το δούμε σήμερα το απόγευμα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω όπως και να έχει είναι ότι η πολιτική συνοχή ε, αποτελεί τμήμα μεν της στρατηγικής για 2020 αλλά είναι και δε ανεξάρτητη από τη στρατηγική αυτή γιατί πληρεί περισσότερους στόχους. Έτσι λοιπόν ε, ήθελα να της δώσω μια διαφορετική διάσταση. Αν ε, και κατανοώ ότι είπε η Πρόεδρος Δηλαδή, αν θέλουμε μία δομή που να επισέρχει μεγαλύτερη ευελιξία, αντί να μιλάμε για εξωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, καλύτερα είναι να τα βλέπουμε πιο καθολικά τα πράγματα. Όμως, θα διαμαρτύρονταν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ραγκή τώρα. Για την εκπαίδευση και την νεολαία, το αναφέρω στον παράγραφο για την ηθαγένεια. Ξεκάσαμε όμως να βάλουμε τη θεματική πρωτοβουλία Youth on Move. λένε κινήσει. Ίσως θα ήταν απαραίτητη μια τέτοια συμπερίληψη. Αλλά βλέπετε, γι' αυτό και συζητάμε, για να βλέπουμε τι λάθη διαπράξαμε όταν εκπονήσαμε την έκθεση και να τα διορθώσουμε μέσω τροπολογιών. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε, έχουμε 12 λεπτά στην διάθεσή μας, περνάμε στο τέταρτο τμήμα της δεύτερης φάσης. Για την τρέχουσα κατηγορία 3 και 4, Θαγένεια και η παγκόσμια Ευρώπη. Στον κατάλογο μιλητών η εξή. Ένας ομιλητής μάλλον. Α, μάλιστα δύο. Α, μα Πολύ ωραία. Αν δεν ε, ολοκληρωθεί το θέμα αυτό σήμερα το πρωί, μπορούμε φυσικά να συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα. Καταρχάς, εισαγωγικά, ο Σαλβαδόρ να μας παρουσιάσει το θέμα. Φεν, Μπέγκε, Φρανσουάλ Φονσί. Και θα δούμε. Παρακαλώ, Σαλβαδόρ. Ναι, Πρόεδρε, πολύ σύντομα μας μένουν ε, τα τμήματα ηθαγενείας ε, και της ε, Ευρώπης στον κόσμο. Βλέπετε για την ηθαγένεια ότι εδώ τα όλα κάτω από τον ίδιο τίτλο. Και εδώ συμπεριλαμβάνω αφενός την ενίσχυση, την προγωγή της ε, ε, ποικιλομορφίας, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, αναφέρομαι και στους νέους και ότι οι πολιτικές για τους νέους και τον πολιτισμό κρατούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 για το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε ολοκληρωμένη εστίαση στα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου. Και ακόμη και αν λαμβάνουν ε, πολύ μικρή χρηματοδότηση, υπάρχει ιδιαίτερη προσθέμενη αξία στις αυτόνομες δημοσιονομικές προοπτικές, στις σημερινές και στις μελλοντικές, γιατί επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν μπορούν να τις διαχειριστούν με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν αφήναμε τα θέματα αυτά να τα διαχειριστούν τα κράτη-μέλη με τα θέματα μεταναστασίας και ασύλου, θα υπήρχαν ε, κράτη-μέλη που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Όλοι γνωρίζουμε έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει καλή χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό, γιατί αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της ευρωπαϊκής σταθερότητας στο μέλλον. Και έχουμε και το θέμα του σεβασμό των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Εδώ δεν έχω συμπεριλάβει κάποια από τα συμπεράσματα που πρότεινε η κυρία Μάλστρουμ ε, στο Στρασβούργο της Ουράλης, γιατί δεν προλάβαμε. Φυσικά συμφωνώ, όμως υπόθηκαν. Και θα υπάρξουν ε, τροπολογίες σχετικά για την Ευρώπη στον κόσμο. Πρώην κατηγορία 4 εξωτερικών δράσεων. Κοιτάξτε, ποτέ δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα στις δημοσιονομικές προοπτικές και στον αντίστοιχο προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε όλες τις αναγκαιότητες παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι ο κύριος ε, χορηγός διεθνούς βοήθειας, αλλά ποτέ δεν θα αρκεί. Έτσι λοιπόν πάντοτε πρέπει να θέτουμε προτεραιότητες, πάντοτε υπάρχει χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών μας των δεσμεύσεων της Κομισιόν του Συμβουλίου και όπιν του τρόπου ερμηνείας ε, στην κατηγορία 4. Υπήρξε η υποχρηματοδότηση χρόνια και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς ευελιξίας για να το αποφύγουμε. Τώρα, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Οι αθώοι τη Επιτροπή Προβλησμού συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε το εξή, ότι αυτό θα αναλυθεί μέσω από τις αρχές αποτελεσματικότητα και πρέπει να αναζητήσουμε την ουδετερότητα του προπολογισμού. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον προπολογισμό ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, αν γνωρίζετε ότι δεν θα το πετύχουμε αυτό. Και κατόπιν υπενθυμίζουμε στην έκθεση τη ε, δεσμεύση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους της χιλιετίας που δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και χρειάζεται ένα πολύ σημαντικό τμήμα των εθνικών προϋπολογισμών και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επίσης, κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στις καταστάσεις κρίσης. Και εδώ με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες στην πολιτική γειτονία. Κυρίως υπό το φως των ανθρωπιστικών κρίσεων που βλέπουμε. Από την άλλη πλευρά της Μεσογείου έχουμε δημοσιονομικό αντίκτυπο μεσοπρόθεσμο. Μιλάμε για τους άμεσους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βλέπετε ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία πολιτικών αλλαγών και θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι προτεραιότητε τη πολιτική γειτονία. Σίγουρα θα υπάρξουν τροπολογίε προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι για το μέλλον πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό κονδύλι. Επίση, γνωρίζουμε ότι ο τρόπο αντιμετώπιση αυτών των ανθρωπιστικών κρίσεων μέσω του μέσου για την ανθρωπιστική βοήθεια και του έκτακτου αποθεματικού είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμός γιατί το αποθεματικό για τις ε, καταστάσεις της επίγουσης ε, για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται να αναλυφθεί ε, πολιτική, να γίνει πολιτικό συντονισμός πρώτα και πολλές φορές δεν μας στάνει ο χρόνος. Η Αρμόδια Επίτροπος άρχισε τη διαδικασία για την ενεργοποίηση, γιατί το αποθεματικό για τη Βόρεια Αφρική και μάλλον θα ξεκινήσει η δικασία 1η Απριλίου. Ξέρετε, εμείς πρέπει να επιμένουμε για μια ταχύτερη ενεργοποίηση αυτού του παθηματικού όταν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά κυρίως αναφέρονται στους ε, τομείς που αφορούν την Ιθαγένεια και την Ευρώπη. Στον κόσμο εδώ δεν ζητούμε αύξηση της χρηματοδότησης, αλλά φυσικά μέσω της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της βελτίωσης των μέσων μπορούμε να βελτιώσουμε τα μάλα τον αποτελεσματικό τους χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητά τους στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Ε, τελειώνει η ώρα μας. Δεν θα προσπαθήσουμε να μιλήσουν όλοι οι ομιλητέ, αλλά θα τα πούμε άλλωστε και σήμερα το απόγευμα, να ξεκινήσουμε με τον Γιώραν, μετά να συνεχίσουμε με τον Ράιμερ, μετά την Φρανσουά, να ακούσουμε και μετά θα κλείσουμε. Άρα, καλό διάλειμμα και τα λέμε στις τρει. Bitte? Ja. Das ist wahr. Das, das macht ja nichts. Das wäre So.